Dobrý dámy Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής μας για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας και να σας πω πως θα μιλήσω τη μετρική μου που είναι βέβαια η τσεχική. Μια και με τον τρόπο αυτό θα μπορώ να εκφραστώ πιο εύκολα. Να σας υπενθυμίσω πως Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να σας υπενθυμίσω. Καταρχήν ότι γίνεται αυτή τη στιγμή ε, web streaming και επίσης πώς καταγράφεται η συζήτησή μας. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, μπορώ να θεωρήσω πως έχουμε εγκρίνει τις ημερήσιες διάταξης. Βλέπω λοιπόν πως δεν υπάρχουν διαιρήσεις, δεν σηκώνει κανείς το χέρι του, εγκρίνεται και μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα σημεία. Για το σημείο 4, για τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας στα πλαίσια της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, να σας πω πως για το σημείο αυτό έχουμε προβλέψει να γίνει και μια ανταλλαγή απόψεων με τον καθηγητή ε, κύριο Λουίς Σιμών που είναι καθηγητής στο ε, Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και ο λόγος για τον οποίο θα συζητήσουμε το σημείο αυτό ε, έχει να κάνει με το σχέδιο έκθεσης που κάνουμε αυτή τη στιγμή που είναι ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις για ε, τη συνθήκη από την κοινή αυτή πολιτική άμυνας και τι ακριβώς ε, ισχύει μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε τον κύριο Γκάλης και τον κύριο Γκονσάλες που έχουν παρουσιάσει ε, το σχέδιο έκθεσης. Έχουμε κάνει και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να καλωσορίσω τον καθηγητή κύριο Λουί Σιμών από, το, ε, τη Σχολή Ευρωπαϊκών Μελετών του ε, Πανεπιστημίου των Βρυξελών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή που μου απευθύνεται. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και πρέπει να σας πω ότι περιμένω με χαρά και τις δικές σας παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ε, κατανοώ κύριε Πρόεδρε πως αυτή τη στιγμή κλείνει μια έκθεση για τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας στα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την άμυνα και τις σχετικές κοινέ ευρωπαϊκές πολιτικές. Και επίσης ε, θέλετε να δείτε πιο συγκεκριμένα κάποιους μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα τη μόνιμη δομή συνεργασίας ή ε, τις μάχημες μονάδες ή το πώς θα γίνει τη χρηματοδότηση των μονάδων αυτών και επίσης και κάποια καυτά πολιτικά θέματα, ε, πώς μπορούμε να έχουμε λοιπόν αυτά τα στρατηγία, τη στρατηγική διοίκηση και πού θα εδρεύει αυτή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε στα συγκεκριμένα σημεία κατά τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα καταρχήν να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να μοιραστώ μαζί σας κάποιους από τους πιο βασικούς στρατηγικούς και πολιτικούς στόχους και ζητήματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν ε, για θέματα ευρωπαϊκής άμυνα στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι το πιο εύκολο για μας είναι ε, να μπούμε σε ένα τέλμα τέρμων νομικών συζητήσεων και να χάσουμε πια ε, από ε, και να απολέσουμε μάλλον τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας, γιατί ξέρετε πως οι στόχοι που έχουμε θεσπίσει πολλές φορές έχουν να κάνουν με ε, ζητήματα που απορρέουν από νομικές συζητήσεις που γίνονται σε, κάποια, σε κάποιους χώρους και λιγότερο από γεωπολιτικά ζητήματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν. Να ξεκινήσω λοιπόν με κάποιες γενικές σκέψεις για κάποια αλληλένδετα θέματα και τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εθνικής Καταρχήν, σε τι είδους στρατηγικές προκλήσεις ε, κινείται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Δεύτερον, ε, πόσο φιλόδοξοι πρέπει να είμαστε σε στρατηγικό επίπεδο και τι είδου στρατηγική ικανότητα χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Και τρίτον, πώς αυτή η κοινή πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί στα παραπάνω ζητήματα. Για την πρώτη ερώτηση που έκανα, δηλαδή τι είδους προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να σας πω πως στα πλαίσια της ε, ε, σφαιρικής στρατηγικής, του Global Strategy, έχουν δοθεί κάποιες πρώτες αποκρίσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί οποιαδήποτε συζήτηση που θα γίνει για το επίπεδο της στρατιωτικής φιλοδοξίας ή για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε στρατιωτική ικανότητα ή για το τι θα γίνει για το μέλλον της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, να σας πω πως θα πρέπει εδώ να ξεκινήσουμε μάλλον ε, προσπαθώντας να δούμε ποιες είναι οι γεωγραφικές και οι επιχειρησιακές παράμετροι τους οποίους θέλει να ακολουθήσει η Ευρώπη στρατηγικές που θεσπίζει. Για την στρατηγική για το 2016, να σας πω ότι εντοπίζει την άμεση γειτονιά ως χώρο προτεραιότητας, στρατηγικής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως ισχύει πως η Ευρώπη αναγνωρίζει πως το περιβάλλον ασφάλεια στην Ευρώπη και στην άμεση ε, γειτονιά της σχετίζεται με το τι γίνεται πιο μακριά. Δηλαδή, στην Global Strategy, για παράδειγμα, αναφέρουμε πώς θα συμμετέχουμε στην ασφάλεια, στα θαλάσσια ασφάλεια, τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια, λόγω των όσων συνέβησαν στον Ειδικό Ωκεανό και στη Μεσόγειο και θα διερευνήσει ε, το τι γίνεται ε, στα στενά της ε, Μάλακα ή στην νότια θάλασσα της Κίνας ή επίσης και στον κόλπο της Γουινέας. Αλλά καταλαβαίνουμε πως όλα αυτά που γίνονται ευρύτερα επηρεάζουν το τι γίνεται στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Οπότε υπάρχει ένα στοιχείο κλειδί στη συζήτηση που είναι η παγκόσμια διάσταση. Όμως, Όμω, και αυτό πρέπει να το τονίσω, παρόλε από τις εξαιρεσει αυτές που σα ανέφερα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ή τουλάχιστον τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη εξετάζουν το τι γίνεται σε απομακρυσμένες περιοχές, το αντιμετωπίζουν κυρίως βλέποντάς το σαν θέμα οικονομικό-διπλωματικό και δεν το βλέπουν από την οπτική γωνιά τόσο πολύ την επιχειρησιακή, τη στρατιωτική ή ακόμα και την καθαρά αμυντική. Οπότε οι συζητήσεις που γίνονται για την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το ΝΑΤΟ και θα το πω αυτό αργότερα, συζητάμε δύο βασικά ζητήματα. Καταρχήν, αποτροπή και να αποφύγουμε α, τους υβριδικούς πολέμους στα ανατολικά μας και δεύτερον πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στην ασφάλεια που προκύπτουν από τη γειτονιά μας στην ε, Νότια Ευρώπη, δηλαδή το ε, Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική και οι χώρες της υποσαχάρης Αφρικής, ε, όπως επίσης και οι χώρες ε, Σαχίλ. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που έχουμε στο Βορρά και στο Νότο, των όσων συμβαίνουν στο Βορρά και στο Νότο και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ενισχύει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά παράλληλα και το ΝΑΤΟ και για τις ε, γεωγραφικές παραμέτρους που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το ποιο είναι το αναδειγμένο επίπεδο στρατιωτικής φιλοδοξία τη Ευρώπης θα πρέπει να λαμβάνει η υπόψη του την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και την άμεση γειτονιά της ως τα βασικά σημεία αφετηρία. Δηλαδή, να είναι αυτά τα βασικά σημεία αναφορά της ζητήσεις που κάνουμε. Τώρα, για τα επιχειρησιακά, να σας πω πως η κοινή πολιτική της Ευρώπης για θέματα ασφάλειας και άμυνας και εδώ σχετίζεται με τη συζήτηση που θα γίνει σήμερα, συνήθως συνδέεται με, μία, με ε, επιχειρήσεις που γίνονται εκτός, αλλά χαμηλής έντασης και με προκλήσεις τις οποίες εμείς θεωρούμε ε, ε, εσωτερικές εξωτερικευμένε, δηλαδή διαχείριση συνόρων, τρομοκρατία κτλ. Όταν μιλάμε για αποτροπή ή για συλλογική άμυνα, τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν πως σε πολύ ισχυρότερη ε, θέση βρίσκεται το ΝΑΤΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα πρέπει να σου πω ότι αυτό ε, ισχύει και για ε, στρατιωτικέ επιχειρήσει υψηλή ένταση εκτό. Δηλαδή κάποιες εμπειρίες που αποκτήσαμε από τη Λιβύη, από τη Συρία ή από το Μαλί δίνουν την εντύπωση πως όταν το στρατιωτικό διακύβευμα είναι αρκετά υψηλό τότε το ΝΑΤΟ και κάποιες ad αποτελούν τις εναλλακτικές λύσεις που προτιμούν τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα κατέληγα στο συμπέρασμα πως οι επιφυλάξεις των κρατών μελών για ένα πραγματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα πραγματικό αμυντικό ρόλο ή συμμετοχή σε ε, υψηλής έντασης επιχειρήσεις ε, εξακολουθούν να μένουν στην επικαιρότητα. Όμως οι επιφυλάξεις αυτές δεν θα έπρεπε να μας παρεμποδίσουν από την δυνατότητα που θα δώσουμε στην κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας έτσι ώστε να αποτελέσει ένα βήμα για συζητήσεις που θα γίνουν για το ποιο θα έπρεπε να είναι το επίπεδο επίπεδο φιλοδοξίες της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ε, ικανότητα ή πολιτική. Γιατί στι συζητήσει αυτές τα κράτη-μέλη θα αποτελέσουν το τελικό σημείο αναφοράς και θα πρέπει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσυπογράφουν ακριβώ τα ίδια κείμενα. Τι σημαίνει αυτό. Να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Γιατί ανεξάρτητα με το αν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα επιλέξουν το χ ή ψ πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, όταν αντιμετωπίσουμε μια πραγματική κρίση και τα πράγματα αγριέψουν, αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη να εξακολουθεί να έχει κάποιο λόγο ύπαρξη, θα πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα που μιλάει το, το ΝΑΤΟ και τα πιο φιλόδοξα κράτη-μέλη σε επίπεδο στρατιωτική ικανότητα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να θέσουμε τον πύχη ψηλά και να σκεφτόμαστε άμυνα, αποτροπή με μεγάλες δυνάμεις, αλλά επίσης και επιχειρήσεις που θα κάνουμε εκτός σε εχθρικά η πολύ στρατιωτικοποιημένα περιβάλλοντα. Και ξέρω ότι αυτή η γλώσσα σοκάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην αισθάνονται άνετα με τέτοιου είδους ε, διατύπωση και δεν λέω αυτή τη στιγμή πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αρχίσει να σκέφτεται ε, πώς μπορεί να κάνει τέτοιου είδους πολεμικές επιχειρήσεις υψηλής έντασης εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ εγώ αυτό να το αποφασίσω, αλλά αυτό που λέω είναι πω είναι σημαντικό η κοινή πολιτική και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν αυτά τα υψηλότερα επίπεδα φιλοδοξία, να ανταποκριθούν, να μπορούν με τον τρόπο αυτό να στηρίξουν τα κράτη-μέλη στι προσπάθειε που κάνουν αυτά για να διατηρήσουν ε, μεγάλη, υψηλή στρατιωτική ε, ικανότητα σαν αυτή που χρειάζεται κανεί σήμερα έτσι ώστε να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδου υψηλή φιλοδοξία. Μιλάμε δηλαδή για επίπεδο φιλοδοξία και κανονικότητα για ικανότητα. Δεν μιλάμε για επιχειρήσεις που θα γίνονται απευθείας μέσω της Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ άμυνας και αποτροπής αφενός και ε, επιχειρήσεων εκτός αφετέρου. Μπορεί κανείς να το ονομάσει όπως θέλει. Ε, Ξέρουμε επίσης πως είναι πολλές διαφορές μεταξύ ε, της ε, ανατολικής ε, γειτονιάς ή σκέλους Ευρω... Ευρώπης και των περιοχών που είναι στο νότο. Αλλά επειδή έχω λίγα λεπτά ακόμα θα προσπαθήσω να δω ακριβώς τι σημαίνουν όλα αυτά και να μπορέσω να ενώσω τις έννοιες βοράς νότος, εκτός, εντός. Δηλαδή Καταρχήν, έχουμε, πολύ, ε, ε, έχουμε οπλικά συστήματα μεγάλης ακριβίας με κατευθυνόμενους και τα κατευθυνόμενα πυραυλικά συστήματα, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Γιατί αυτή τη στιγμή η συζήτηση που κάνουμε θα έπρεπε να έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στον κόσμο σήμερα. Ποια είναι τα βασικά ε, προβλήματα. Και αυτή η διάδοση αυτών των συστημάτων οπλισμών υψηλής ακρίβειας αποτελεί και τη βασικότερη πρόκληση για τους Ευρωπαίους και αυτό ξεπερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γιατί από το τέλος του ψυχρού πολέμου οι περισσότερες ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ε, ε στρατιωτική φιλοδοξία και την στρατιωτική ικανότητα και εδώ μπαίνουμε στον πυρήνα της συζήτησης. Αυτές οι συζητήσεις επαναλαμβάνω από το τέλος του ψυχρού πολέμου γίνονται λαμβάνοντας υπόψη πως ε, κυριαρχεί η δυτική τεχνολογία, ε, η στρατιωτική παγκόσμια. Όμως η παγκοσμιοποίηση ακριβώς έχει σημάνει πως έχουμε μια σταδιακή ε, σταδιακή διάδοση αυτών των ε, πυραυλικών συστημάτων και των κατευθυνόμενων στρατιωτικών και οπλικών συστημάτων σε χώρες που δεν είναι δυτικές Οπότε μιλάμε ε, όχι μόνο για κράτη αλλά και για ομάδες έχουν έτσι ε, δημιουργήσει ε, χώρους στους οποίους εμείς πλέον δεν έχουμε πρόσβαση γιατί έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικού πολέμου, κύβερνου πολέμου, προστασίας μέσω αντιπυραυλικών συστημάτων κτλ. Οπότε όταν μιλάμε για ικανότητα, μιλάμε για ικανότητα που έχει ως σκοπό να αποτρέψει αυτές οι δυνάμεις να μπορούν να επέμβουν σε συγκεκριμένη περιοχή και για ικανότητα που περιορίζει τη δυνατότητα μετακίνησης κάποιων ομάδων από τη στιγμή που βρίσκονται σε συγκεκριμένη πολεμική περιοχή. Πάντως, οι εξελίξεις αυτές με το γεγονός ότι έχουμε αυτή την διάδοση αυτών των ε, τηλεκατευθυνόμενων οπλικών συστημάτων και τις περιοχές στις οποίες πλέον εμείς δεν έχουμε πρόσβαση, έχουμε οδηγηθεί σε έναν κόσμο που πλέον διακυβεύεται η, η τεχνολογική κυριαρχία του δυτικού κόσμου. Την περασμένη δεκαετία οι περισσότερες συζητήσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό της διάδοσης έγιναν στα πλαίσια ε, του κινέζικο-αμερικανικού πολεμικού ανταγωνισμού στο δυτικό ειρηνικό. Όμως, η διάδοση αυτών των τηλεκατευθυνών οπλικών συστημάτων και των περιοχών μη πρόσβαση δημιουργεί πια σοβαρά προβλήματα και στου Ευρωπαίου. Και τα προβλήματα αυτά έχουν πάρα πολύ σοβαρέ επιπτώσει και στα πλαίσια τη Άμυνα και τη αποτροπή και στου ιδρυδικού πολέμου, όχι μόνο στα ανατολικά μα σύνορα αλλά και σε πολεμικέ επιχειρήσει που θέλουμε να κάνουμε εκτό σύνορα μα στο Νότο. Και για να κλείσω, να σα πω πω τα τελευταία χρόνια η Ρωσία, για παράδειγμα, στα ανατολικά μας έχει καταφέρει να κάνει μεγάλη πρόοδο ε, με τα συστήματα αυτά, οπότε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που είναι ε, όμορες της Ρωσίας ε, πραγματικά είναι τροτές αυτή τη στιγμή και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πληγούν από τέτοιου είδους οπλικά συστήματα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα ε, και στο θεματολόγιο της αποτροπής στην Ευρώπη, γιατί σε περίπτωση σύραξης ή κρίσης είναι πλέον στρατιωτικά πολύ επικίνδυνο οι Ευρωπαίοι να μετακινήσουν είτε στρατεύματα είτε ε, καράβια είτε αεροπλάνα στις περιοχές αυτές τις γειτονικές ε, στον, ε, γειτονα, στα ανατολικά μας σύνορα γιατί ακριβώς ε, υπάρχει κίνδυνος κατά τη διάρκεια αυτών των μετακινήσεων από και τα οπλικά συστήματα αυτά αλλά και το γεγονότος πως δημιουργούνται περιοχές μη πρόσβασης. Πρέπει να σκοπεύω στο το πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο με την Ανατολική Ευρώπη, γιατί αυτό τα τηλεκατευθυνόμενα οπλικά συστήματα ή πυραυλικά συστήματα εξαπλώνονται και προς ε, την διευρυμένη ε, ε, νότια γειτονιά, στη Βόρεια, νότια, στη Βόρεια Αφρική, με στην Ερυθρά θάλασσα, στην, στο Λεβάντε. Οπότε εκεί σε τεχνολογικό επίπεδο η εξέλιξη δεν είναι τόσο ε, μεγάλη, αλλά υπάρχουν κάποιοι κρατικοί φορείς και κάποιες μη κρατικές ομάδες που δημιουργούν αυτή τη στιγμή, που χρησιμοποιούν μάλλον τις ε, ευκαιρίες τεχνολογικές που δίνουν αυτά τα οπλικά συστήματα έτσι ώστε να δημιουργούν τις δικές περιοχές μη πρόσβασης για να μπορούν ε, να δρουν αλεξέλεκτες. Για παράδειγμα, το Ιράν και τα όσα έκανε στα στενά του Ορμούς η Συρία με το σύστημα αντιεροπορικής ε, προστασίας και αυτό που έγιναν στην Ιεμένη με τους Χούτι οι οποίοι χρησιμοποίησαν τηλεκατευθυνόμενους πυράβλους κατά ε, πλοίων ε, για να προστατεύσουν ε, τα δικά του συμφέροντα. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη και για τις ικανότητες στρατιωτικές ε, που πρέπει να αναπτύξουμε και τι σημαίνει για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα. Αλλά από τα τέλη του ψυχρού πολέμου, όπως σας είπα, το δεδομένο πως έχουμε την ελευθερία στρατιωτικής πρόσβασης και μετακίνησης ε, είναι η σκέψη που έχει κατευθύνει την στρατηγική πολιτική που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι περισσότερε ευρωπαϊκέ συζητήσει, σε επίπεδο από τη δεκαετία του 90 και από την ανάπτυξη ανάπτυξη στρατιωτική ικανότητα είτε στο ΝΑΤΟ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε και μέσα σε μεμονωμένα κράτη-μέλη έχουν περιστραφεί γύρω από το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση, πώς μπορούμε να λαμβάνουμε ε, κάποιες αποφάσεις για ειρηνευτικές παρεμβάσεις σε ήρεμα περιβάλλοντα και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που μετά μπορούμε να στείλουμε δυνάμει ταχεία ε, δράση ε, κτλ και μάλιστα από το 2003 και μετά έχουμε το παράδειγμα και των μάχημων μονάδων αλλά ε, και των μονάδων ε, άμεσης απόκρισης ε, που έχουν να κάνουν με το πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να επένδυσει στρατιωτικά ή επιχειρησιακά σε μια συγκεκριμένη σύραξη. Εμείς δηλαδή έχουμε δώσει ε, προτεραιότητα στις ε, επικοινωνίες ε, μέσω δορυφόρων ή στον ανεφοδιασμό αεροπλάνων στον αέρα και όχι τόσο πολύ σε κάποιες άλλες ικανότητες που θα έπρεπε να έχουμε αναπτύξει γιατί μιλάμε για πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι stealth, είναι πολύ βαριές, είναι πολύ ορατές και οι οποίες είναι πολύ τρωτές σε κάποιο είδους ε, τηλεκατευθυνόμενη ε, επίθεση. Και για τον τρόπο αυτό, για τον λόγο αυτό θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι να σκεφτούν περισσότερο το τι πρέπει να κάνουν με την τεχνολογία τους, έτσι ώστε η τεχνολογία που θα επιλέξουν να μπορούν και σε ένα αρνητικό περιβάλλον μη πρόσβαση να φανούν αποτελεσματικές. Για τις συζητήσεις που έχουν γίνει για το πόσο φιλόδοξοι πρέπει να είμαστε για τα τελευταία 30 χρόνια σε στρατιωτικό επίπεδο, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να κριθούν ως λανθασμένες στην οπτική γωνία που έχουν ακολουθήσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τεχνολογίες και στρατιωτική ικανότητα που θα μπορούν να μας επιτρέψουν να δράσουμε σε όρημα περιβάλλοντα μη πρόσβασης έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να είναι αποτελεσματικοί γιατί οι ανταγωνιστές μας σήμερα και στο μέλλον μάλλον θα έχουν, το ίδιο, ε, θα έχουν τα ίδια συστήματα ε, απόλυτης ακρίβειας τηλεκατευθυνόμενα ε, οπλικά ή πυραυλικά ακριβώς τα ίδια που έχουμε κι εμείς. Οπότε όταν λέω εμείς ενώ εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό και πριν κλείσω... Γιατί πρέπει να δούμε και το τι ακριβώς θα συμβεί με τους μηχανισμούς που έχουμε στην ε, διάθεσή μας και με τους διάφορα ε, θεσμούς που αποτελούν τα κομμάτια της κοινή ε, πολιτικής. Να πω λοιπόν, και νομίζω είναι σημαντικό να ξανατονιστεί αυτό, πως οι Ευρωπαϊκέ και οι Διατλαντικέ συζητήσει για το επίπεδο φιλοδοξίας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που προκύπτει συνέχεια, και την στρατηγική ικανότητα που θα εξελίξουμε, να δεχτούμε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο ε, μοντέλο ε, στον κόσμο, στρατιωτικό, που έχει να κάνει με την παγκόσμια διάδοση οπλικών συστημάτων ακρίβεια τηλεκατευθυνωμένων, το και ε, περιεχών μη πρόσβασης. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι Ευρωπαίοι για να τα καταλάβουν όλα αυτά να διερευνήσουν και τα κανάλια που έχουν ε, επικοινωνίας που είναι διμερή αλλά και όλα τα πολυμερή και να δούνε το θέμα της τεχνολογίας και της τεχνολογικής καινοτομίας κάτι στο οποίο έχουν προχωρήσει περισσότερο οι ΙΠΑ για παράδειγμα τεχνολογική στρατιωτική καινοτομία και όπως αυτή στηρίζεται και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και άλλες πληροφορίες όμως ένα τελευταίο δεδομένο των προοπτικών πως αυτή τη στιγμή στην διαδικασία που τρέχει στο ΝΑΤΟ θα πούμε πως ε, για το σχεδιασμό των δομών, ε, των στρατιωτικών δομών στην Ευρώπη ακολουθεί ε, την πάγια τακτική, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να λάβουμε υπόψη και το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ τουλάχιστον στο σχεδιασμό ικανότητας να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Περισσότερες προσπάθειες λοιπόν για να συνδέσουμε και το διεθνές ε, και το διεθνές προσωπικό του ΝΑΤΟ και το ΣΕΙΠ με, ε, τις, ε, με τους ομολόγους του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια και τα αρχηγεία και τη στρατιωτική και στρατηγική διοίκηση του ΝΑΤΟ να τη συνδέσουμε με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοικήσεις έτσι ώστε το επίπεδο ικανότητας και φιλοδοξίας να είναι παρόμοιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δεν θα πω άλλο. Σας ευχαριστούμε καθηγητά. πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που επισημάνατε εσείς στην παρουσίασή σας. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να επέλθει μια εξισορρόπηση ανάμεσα στον Νότο και την Ανατολή Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει διαίρεση ακόμη και στο Κοινοβούλιο. Δύο μεγάλες κατηγορίες. Από τις επωνομαζόμενες παλιές χώρες, όλοι οι βουλευτές που είναι από τις επωνομαζόμενες παλιές χώρες και όλοι που έρχονται από τις νέες χώρες που ανήκαν στο Σοβιετικό μπλοκ. Όσοι από εμάς Είχαμε εμπειρία σε σχέση με την εισβολή από την Ανατολή. Μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανησυχίες των παλιών χρόνων όπως της Ισπανίας για την εισβολή από τον Νότο. Για τα στρατηγικά ζητήματα νομίζω θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς στη λευκή βίβλο για την άμυνα Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε για τον επιμερισμό ε, των ε, καθηκόντων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Έχετε πιο συγκεκριμένες ιδέες για τα αμυντικά ζητήματα, πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτός ο επιμερισμός, κυρίως για τις αμυντικές προσπάθειες. Αυτή είναι η προσωπική μου ερώτηση. Ταυτόχρονα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στην κύριο Χάν. Ε, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Καθυστέρησε η πτήση μου. Πρόλαβα το τέλος της παρουσίασής σας, δυστυχώς. Μόνο θέλω ε, να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε για την τρομοκρατία. και την ε, κοινή αντίληψη περί τρομοκρατίας. Είναι σαφές ότι είναι πηγή ανησυχία για μας και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Και ως εκ τούτου χρειάζεται συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. κάντας μια ε, αναδρομή όμως βλέπουμε ότι πηγάζουν αυτά τα φαινόμενα, αυτή η αλυσίδα από τους ε, μαχητές της ελευθερίας που μετά έγιναν ε, Ταλιμπάν, μετά έγιναν στο τέλος αλτάες. δεν υπάρχει μια αλυσίδα, μια αλληλουχία. Υπάρχει τρόπος να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα, όπως πρέπει να το εξετάσουμε από διαφορετικό πρίσμα. Το δεύτερο που αναφέρατε είναι τα καθοδηγούμενα πυρομαχικά ακριβίας. Και μιλήσατε για την Ιεμένη και τους ε, Χούτι. Για πιθανή χρήση αυτών των πυρομαχικών. Ε. Και ε, αν δούμε και το Ιράν και τις ναυτικές βάσεις που προσπαθούν να έχουν, μεταξύ άλλων και στην Ιεμένη, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν συμβεί αυτό. Ε, τώρα, για την άποψη της Ευρώπης, εξελέγει ο Ντόναλτ Τραμπ. Έχουμε την ε, άλλη υπερδύναμη με τον ε, επιθετικό Πούτιν που με πυγμή διεκδικεί ε, κομμάτια της Μέσης Ανατολής, στη Συρία παραδείγματος χάρη. Αν τώρα δούμε και στρατιωτικές ασκήσεις στο Πακιστάν και την Κίνα, ποιες ε, επιπτώσεις έχουν αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Σάιμον, ε, σας ευχαριστούμε για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις σας. Πρόεδρε. Με ενέπνευσε και εμένα ο κύριος Σάιμον, όπως και εσάς. Για να αρχίσω την ε, παρέμβασή μου με ένα κοινό τόπο ουσιαστικά. Έχουμε ε, ε, την εντύπωση όπως οι άλλοι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό όραμα πίσω από την κοινή πολιτική. Με την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση και την πίεση της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ομοψυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Οι χώρε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δεν αναγνωρίζουν τι απειλέ ασφάλεια που αντιμετωπίζουν ε, οι χώρε του Νότου. Υπάρχουν ε, διαχωριστικές γραμμέ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξίσου σημαντικέ κατά τη γνώμη όσο και πιέσει έξωθεν όταν μιλάμε για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Κύριε καθηγητά, δύο ερωτήσεις. Άρθρο 42, εδάφιο 7 τη συνθήκη Λειτουργίας της Ένωσης. Πώς να αποφύγουμε την ε, παρανόηση, θα θυμάστε με τις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι, πρώτη φορά επικαλέστηκε αυτό το άρθρο της συνθήκης ένα κράτος μέλος. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε την κίνηση της Γαλλίας και πώς να μην παρεμηνευτεί αυτό το άρθρο. Δεύτερον, για τα ευρωπαϊκά σύνορα και την ακτοφυλακή. Ξέρετε, το Σεπτέμβρη του 2016 ε, δόθηκε το πράσινο φως από το Συμβούλιο. Ποια είναι η απόψή σας Δοθή τη κατάσταση είναι η προσφορότερη προσέγγιση. Εφόσον μιλάμε για κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα, ή κατά περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, διότι η συνορία φυλακή και ακτοφυλακή ενδεχομένως να συνιστούν απαντήσεις στις τρέχουσες απειλές και σε πολιτικά φαινόμενα που ε, οδηγούν σε κλειδονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνταράσσουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Έχω εγώ όμως άλλη μια ερώτηση. Η κίνδυνοι εξ Ανατολής, όταν μιλάμε για την Βαλτική, για την Πολωνία. Ε, γιατί μην ξεχνάμε ο, ότι υπάρχει περιοχή ε, του Καλίνιγκρετ με τους πυράβλους, ε, με ε, τόσο μεγάλη εμβέλεια που μπορούν να πλήξουν ε, όλες τις ε, πρωτεύουσες των χωρών της Βαλτικής και την Βαρσοβία. Γιατί έχουν 500 χιλιόμετρα εμβέλεια πια. Είναι η άποψή σας για το άρθρο 5 της συμφωνίας αμοιβαίας προστασίας Θεωρείται ότι στην περίπτωση της Βαλτικής πληρούνται οι προϋποθέσεις ε, για ε, να επικαλεστεί μια χώρα το άρθρο 5 της ε, Διατλαντικής Συμφωνίας. So, Απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Πολύ εύστοχα τα ερωτήματά σας. Θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω, διότι υπάρχουν κοινά ζητήματα. Ε, αρχίζω με το τελευταίο με το οπλικό σύστημα Iskander χρειάζεται πολιτική απόφαση για να ε, κινητοποιηθεί το άρθρο και για να χρησιμοποιηθεί το άρθρο και χρειάζεται σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Για αυτές τις ε, ε υβριδικές, ε, όπως ονομάζονται, απειλές, ε, είναι θεμητό το ερώτημα και θεμητές οι ανησυχίες, διότι οι απειλές ε, στο ανατολικό μέτωπο είναι απειλές ε, κάτω από τη ζώνη, όπως θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε, και όχι παραδοσιακές, ε, καθαρές στρατιωτικές σειράξεις δηλαδή. Ξέρετε ότι και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και στη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούμε πολύ τους υπηρετικούς πολέμους και το συνδυασμό διαφόρων μηχανισμών, διαφόρων μέσων π.χ. χρήση ενεργειακής πολιτικής ε, για την άσκηση πίεσης, ε, το, το τοπικό σύστημα Ισκάντερ, ε. και ούτω καθεξής. Είναι ένα είδος ψυχολογικού πολέμου που ενισχύεται από, τη... από το στρατιωτικό συσχετισμό δυνάμεων με τη Ρωσία. Ε, αναφερθήκατε στο Καλίνιγκρα και τους πυράβλους που έχουν κατασταθεί εκεί. Όταν ε, μιλούσα για τη δυναμικότητα στην Ανατολή, για την απαγόρευση πρόσβασης και αποκλεισμού από περιοχές, Ε, υπάρχουν οι ναι, πυραυλοί ε, ε, βραχές που καλύπτουν ούτως ή άλλως ε, τις χώρες της ε, Βαλτικής ε, και χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, Σουηδία, Φινλανδία. Με αυτά τα ε, πυραυλικά συστήματα ε, απαγόρευσης πρόσβασης στο ανατολικό μέτωπο Καλίνιγραν, Νόρμανς, ε, στο ε, Σεβαστούπολη, στην ε, Κρυμαία. Ε, δημιουργείται δηλαδή μια φυσαλίδα απαγόρευση της πρόσβασης στον εύξηνο πόντο, έτσι την ονόμασαν ε, κάποιοι επιτελάρχες. Και στη Συρία σε σχέση με τις ρωσικές ε, στρατιωτικές βάσεις και αυτό που με ρωτήσατε για το Ιράν που θέλει να ανοίξει ναυτικές βάσεις αλλού ε, και ότι έχει δυναμικότητα απαγόρευσης πρόσβασης και αποκλεισμού. Ε, λοιπόν, δημιουργείται ένα επιχειρησιακό πρόβλημα, αλλά και πολιτικό για τους Ευρωπαίους, διότι η πολιτική και διπλωματική επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε είναι συνάρτηση μιας ε, στρατιωτικής ισορροπίας. Ε, μπορεί να έχουμε πολιτικές πρωτοβουλίε που διατυπώνται με ευρωπαϊκού όρου ε, και με ευρωπαϊκά πρότυπα. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε, διότι υπάρχει μια στρατιωτική υπερδομή που είναι υπέρμα ημών. Και αυτό θα έλεγα ότι ισχύει και για την Ανατολή και για τον Νότο ξυπακούεται ότι ισχύουν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Το πρόβλημα της εξάπλωσης των πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων ακριβίας είναι ένα πραγματικό ουσιαστικό πρόβλημα. Στο Νότο και το Ιράν μάλλον εξαίρεση είναι, διότι σε σχέση ε, με τα πάλι των ανταγωνιστών είναι ιδιαίτερα προηγμένο. Με την εξαίρεση του Ιράν που βρίσκεται σε πολύ ε, προεκχωρημένο στάδιο, για τις επιθέσεις. Ε, στον Νότο θα το χαρακτήριζε αυτό το πρόβλημα μάλλον μελλοντικό, παρότι σε κάποιο βαθμό υφίσταται και τώρα. Και η Συρία έχει πολύ πυκνό ε, δίκτυο αεροπορικής άμυνας και η Εμένη, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή. Νομίζω ότι επανερχόμαστε και στο προηγούμενο ερώτημά σας για τον επιμερισμό των καθηκόντων και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνα, διότι κάποιοι αναφερθήκατε στη Λευκή Βίβλο. Θα μας βοηθούσε αυτό να συνειδητοποιήσουμε για τι πράγμα μιλάμε για το περιβάλλον των απειλών που δεχόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχουν πολύ καλύτερε επιδόσεις σε σχέση με την ενεολογική προσέγγιση των απειλών από τον Νότο, ε, ούτως ώστε να αριοθετήσουν τους ε, κινδύνους που διαπιστώνονται σε αυτή την περιοχή. Ε, με ρωτήσατε για το άρθρο 42.7 για την άμυνα και την αποτροπή. Δημιουργείται πολύ μεγάλη σύγχυση σε τέτοιου είδου συζητήσει που είναι πολιτικά εξαιρετικά φορτισμένε. Νομίζω, το ξεκαθαρίσατε κι εσείς, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον νομικά και νεολογικά εξακολουθεί να υπεραμείνεται της, ε, τη συλλογική άμυνα για την αναχέτηση και για τις επιχειρήσεις υψηλής συχνότητας οι περισσότερες επιχειρήσεις βάσει κοινή πολιτικής ήταν ε, μάλλον στα χαμηλά επίπεδα της πυραμίδας ως προς την ένταση των επιχειρήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, αποκλείονται ε, επιχειρήσεις στα πλαίσια των αποστολών του Πίτερσπεκ, παραδείγματος χάρη για ειρηνευτικού σκοπούς, ε, να αναλυθούν και επιχειρήσεις σε υψηλή ένταση. Γι' αυτό πολιτικά και ενοιολογικά για την άμυνα και την αποτροπή αλλά και για τις επιχειρήσεις εκτός πεδίου ε, υψηλής έντασης. Υπάρχει αυτή η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, θα εξακολουθήσει να υπάρχει και ε, δεδομένων των εξελίξεων. Ε, έχει νόημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει σάρκα και οστά σε αυτή την δέσμευση που έχει αναλάβει διότι Ξέρουμε ότι στις ευρωπαϊκές συζητήσεις στρατηγικού χαρακτήρα αυτό είναι στοιχείο κλειδί για να διατηρήσει λοιπόν το κύρος και τη σημασία της η Ευρωπαϊκή Ένωση ω ε, αμυντικός φορέας στα μάτια των κρατών μελών θα πρέπει να εμπλακεί και σε ε, συζητήσεις υπεριάμυνας και αποτροπής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να γίνεται παράλληλα αυτό στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν συζητήσεις για το επίπεδο φιλοδοξίας ε, και την ανάπτυξη δυναμικότητας και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι στο ίδιο μήκο κύματο η Ένωση και το ΝΑΤΟ και μια διαφορετική συζήτηση το ποιος κάνει τι σε επίπεδο επιχείρησης. Αυτό αφορά τα κράτη-μέλη. Σε παγκόσμιο επίπεδο η στρατηγική επιβάλλει ετοιμότητα για την άμυνα για την προστασία την αποτροπή εξωτερικών απειλών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα προκρίνουν τον ΝΑΤΟ ή άλλου είδους συμμαχίες όταν ε, δημιουργηθεί πρακτική ανάγκη, ε, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ και κυρίως με τα κράτη-μέλη της για την ε, ε, στρατιωτική ικανότητα που θέλει να αναπτύξει. Για το σχέδιο υλοποίηση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες βλέπουμε ότι καταργείται κάθε μία στην αποτροπή. Αυτό είναι ατυχές. Αυτό υπερβαίνει και το πεδίο πραγματογνωμοσύνης μου, γιατί με ρωτήσατε για την τρομοκρατία, τη συνοριοφυλακή και εκτοφυλακή. Ε, πάντως, ε, στη νότια γειτονία οι περισσότερες απειλές δεν συνδέονται με πραγματικές στρατιωτικές προκλήσεις και απαιτούνται μάλλον πολιτικές λύσεις και ε, λειτουργίες ε, μάλλον αστυνόμευσης ε, και όχι επιχειρήσεων υψηλή ένταση. Θα σταματήσω εδώ. Α, ένα λεπτό γιατί θυμήθηκα, με ρωτήσατε και για τον Τραμπ. Ας μην προτρέχουμε και προδικάζουμε τι σημαίνει η εκλογή του. Στον τομέα τη εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα ε, ε, ε, ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διορισμοί που θα κάνει και που έχει ήδη κάνει σε ένα ορισμένο σημείο. Κυκλοφορούν όλε αυτέ οι φήμε και ιστορίε για το πόσο κολλητό είναι με τον Πούτιν και τι θα κάνει σε σχέση με την Ρωσία νομίζω πως θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε αυτά που είπε στην ε, προεκλογική του εκστρατεία και σε αυτά που όντως θα κάνει. Όχι ότι άλλα έλεγε και άλλα θα κάνει, αλλά σκέφτεται να κάνει, αλλά γιατί φιλτράρονται αυτά που λέει από το σύστημα και ε, στο Κογκρέσο θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη για να πετύχει αυτά που υποσχέθηκε ότι θα κάνει για τις διατλαντικές σχέσεις ήταν ε, αρκετά ε, αμφίροπος ο λόγος του ε, και το αφήγημά του μπορούσε να οδηγήσει σε επιχείρους τίτλους, αλλά είναι αρκετά ε, αφήσω ο να για να μπορέσει να πάει προς διάφορες κατευθύνσει, και μάλλον ήμουν και εγώ αφήσω τώρα στην απάντηση που έδωσα, αλλά θα σταματήσω.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

total territory of Nainawa province that ISIS captured during its ε, ε, που είχε καταλάβει ο ISIS μέχρι το 2014 ε, βάσει αμερικανικών πηγών το 25% της Μουσούλης ανακατακτήθηκε από Ιρακινά στρατεύματα τα οποία έχουν αξιοσημείωτες στρατιωτικές επιτυχίες. Σίγουρα όμως δεν έχει λήξει η σύραξη και ε, σίγουρα θα είναι παραταταμένος και αιματηρός ο πόλεμος ε, με πάρα πολύ ε, σοβαρές επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι το αποτέλεσμα ίσως να καθορίσει το μέλλον του Ιράκ. Υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις αλλά και πολιτικά προβλήματα εν Τα στρατιωτικά εμπόδια έχουν ως εξής. Αρχικά, οι δυνάμεις του Ιράκ αντιμετωπίσουν ένα παράδοξο καθώς γίνεται πιο έντονη η μάχη κατά του ε, ISIS. Όσο πιο πολλές περιοχές απελευθερώνουν, τόσο πιο κοντά φτάνουν στο ε, επίκεντρο του ISIS, το οποίο είναι το δυτικό κομμάτι της πόλης Μουσούλης αλλά και το Ταλάφερ και έχουν να αντιμετωπίσουν έναν έξυπνο βίο εχθρό που ξέρει να προσαρμόζεται σε μια πόλη όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύρια ε, άμαχοι, το οποίο είναι μια μεγάλη πρόκληση για οποιοδήποτε στρατό του πλανήτη. Αυτό επιβραδύνει ε, την πρόοδο των μαχητών κατά του ISIS ε, και δυσχεραίνει την ανάκτηση περιοχών. Ε, διότι ε, γίνονται μάχες ε, πόρτα με πόρτα και πρέπει να προσέχουν ώστε να μην βλάψουν αμαχούς πολίτες. Δεύτερον, η πόλη της Μουσούλης αυτή τη στιγμή έχει περικληρωθεί από τα ανατολικά, τα βόρεια και τα νότια. Αυτό, αυτό περιορίζει την κίνηση του ISIS εντός και εκτός της πόλης και περιορίζει επίσης τον ανεφοδιασμό ε, του ΑΕΣΙΣ από το υπόλοιπο της χώρας ε, καθώς επίσης και από άλλες περιοχές της Συρίας. Η Τυράκα συγκεκριμένα όμως το ISIS συνεχίζει ε, να ελέγχει τα 60 χιλιόμετρα διαδρομής που βρίσκονται μεταξύ της Μουσούλης και της πόλης Ταλάφαρ, όπως επίσης και την ίδια αυτή πόλη. Αυτά λοιπόν ε, εμποδίζουν από το να περικυκλώσουν την πόλη από τα ε, δυτικά. Επίσης, ε, ο ISIS χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Οι στρατιώτες του Άισις μετακινούνται μέσα, σε, μέσα από τούνελ στην πόλη, χρησιμοποιούν αυτοκίνητα τα οποία περιέχουν εκρηκτικά και χρησιμοποιούν ελεύθερους σκοπευτές. Επίσης υπάρχει ένας κοινό εχθρός αλλά όχι μια κοινή ατζέντα. Είναι ενωμένοι από την οργή που έχουν προς τον ISIS όλα τα στρατεύματα καθώς επίσης και τα εγκλήματα που, έχουν, που έχει διαπράξει ο ISIS και δικαίως. Όμως ως εκεί φτάνει το θέμα που τους αιωνώνει. Οι, οι θέλουν να καταλάβουν ε, το, την πόλη Αλτάφαρ, ε, οι ε, Πεσμεργά θέλουν να καταλάβουν άλλες περιοχές, το ΠΚΚ θέλει να κρατήσει τον έλεγχο της Σεντζάρ, στρατεύματα των θρησκευτικών μειονοτήτων, γιαζίδιδες, σαπάκες και χαλδαίοι και χριστιανοί θέλουν να τιμωρήσουν τους ντόπιου Σουνίτες πληθυσμούς, τους οποίους θεωρούν ότι συνεργάζονταν με τον ISIS. Αυτή η πολυπλοκότητα στόχων ε, λοιπόν ε, κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη μάχη αλλά και οποιασδήποτε μελλοντικές πολιτικές συμφωνίες. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, μετα-ISIS ε, πολιτική κατάσταση ε, μετά την απελευθέρωση της Πολσούλης. Αρχικά θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι σε περίπτωση που καταληφθεί, απελευθερωθεί η Μουσούλη δεν έχει ιτηθεί ο ISIS. Όπως σε κάθε άλλη περιοχή, όπως το Σαλαχαντίν, Τζιάντ, το ISIS ε, είναι επιτυχημένο όσον αφορά τις ε, παραδοσιακές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των άμαχων αλλά και στρατιωτικών στόχων και αυτή η απειλή λοιπόν δεν θα εξαφανιστεί από τη στιγμή που θα απομακρυνθεί από τη Μουσούλη. Παρά τις ε, στρατιωτικές επιτυχίες, το ISIS αντέχει και έχει την ικανότητα να παραμείνει μια στρατιωτική στρατιωτική οργάνωση. Έχει τη δυνατότητα να δράσει ανεξάρτητα, να πραγματοποιήσει θανάσιμες επιθέσεις όπως συνέβη με το Ισλαμικό κράτος ε, στο Ιράκ ε, μετά την ήττα ε, στη Μουσούλη το Ισλαμικό κράτος θα επιστρέψει στην έρημο οι τεράστιε ερμικές περιοχές ε, μεταξύ Συρίας και Ιράκ είναι ιδανικές ε, για να αποστραφεί, ε, αποτραβηχθεί το ISIS, να βρει καινούριου μαχητέ και να υποφεληθεί από την περιθωροποίηση, την έλλειψη κράτους δικαίου και, την, και τον αποκλεισμό από την πολιτική. Η μάχη της Μοσούλης θα χαρακτηρίσει το μέλλον ε, του Ιράκ, αλλά η μάχη στο Αλάφερ θα χαρακτηρίσει το μέλλον της ε, μάχης. Επίσης υπάρχει η λωρίδα των 60 χιλιόμετρων που φεύγει από τη Μοσούλη. Ε, πριν το 2013 είχε έναν πληθυσμό Τουρκμενίων κυρίως. Το 1 τρίτο ήταν Σουνίτες, 1 τρίτο Σιάτ, ξύν τους Κούρδους. Το 80 λοιπόν ο ε, Χουσέιν τους ε, παραχώρησε γη και ήταν αρκετά περιθωριοποιημένοι. Οι Σουνίτες Τουρκμένοι επίσης ε, την περίοδο του Σαντάμ συμμετείχαν στις δυνάμεις ασφαλείας και μετά την πτώση του καθεστώτος η κατάσταση δυσχεράθηκε, το Ταλάφαρ λοιπόν έγινε ένα προπύργιο για τον Άισις. Σύμφωνα ε, με ε, στοιχεία, με βάση τη στρατηγική του εγκύτητα στη Συρία, το Ταλάφαρ έγινε ένας αυτοκινητόδρομος, ε, αυτοκινητόδρομος για τζιχαντιστές. Το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και τώρα το ISIS. Μετά την κατάληψη από το ISIS το 2014 ε, το ISIS απέβαλε τους Τουρκμένιους ε, και ε, οι μονάδες ιητών κατέλαβαν χωριά και περιοχές και έχουν φτάσει και στην πόλη. Δεκάδες χιλιάδες έχουν φύγει από την πόλη, μερικοί προς τη θάλασσα και στα σύνορα, ενώ άλλοι πηγαίνουν σε περιοχές κατηλημένες από τον ISIS. Οι δράσει λοιπόν των προστρατιωτικών θα καθορίσουν το μέλλον αυτής της πόλης, καθώς επίσης και το μέλλον της επίθεση στη Μοσούλη. Και ίσως να διώξουν τους συνήτες με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα εύπορο έδαφος για, τους, για τον ISIS ώστε να επιστρέψει. Ακόμα και να οδηγήσει μια διαμάχη μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας οι δυνάμεις ασφαλείας ε, αλλά ε, και οι ΣΥΙΤΕΣ θα απελευθερώσουν την πόλη ε, θα επιβάλλουν το κράτος δικαίου και έτσι ίσως να μην έχουμε το χειρότερο σενάριο. Τώρα όσον αφορά τις διαφωνίες, τις εδαφικές διαφωνίες, όλες αυτές θα έρθουν στο προσκήνιο μετά την απελευθέρωση της πόλης. Έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν περιοχές πριν από την απελευθέρωση του Οκτωβρίου, όμως ε, θα συζητήσουν για περιοχές ε, που έχουν απελευθερωθεί μετά την 17η Οκτωβρίου. Για την ώρα οι δυνάμεις των Κούρδων και του Ιράκ αγωνίζονται δίπλα-δίπλα κατά του ISIS, όμως είναι δύσκολο να προβλέψουμε το τι θα συμβεί μετά την ήττα του ISIS. Η πιθανότητα στρατιωτικής ε, διαμάχης είναι πιθανή και με βάση τις θρησκευτικές διαφωνίες δεν είναι γνωστή το ε, ποια σουνητική παράταξη θα ελέγχει την πόλη. Κλείνοντας λοιπόν, ίσως να χρειαστούν μήνες μέχρι να εκδιωχθεί ο Άισις από τη Μοσούλη, όμως το σημαντικότερο ερώτημα είναι το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Η απελευθέρωση της Μοσούλης ίσως να οδηγεί σε μια νέα αρχή για το Ιράκ, αλλά και στη δημιουργία ενός ε, περιεκτικού ε, Ιρακινού κράτους, το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις όρους. Πρώτον, οι αρχές του Ιράκ θα πρέπει να κερδίσουν και πάλι ε, την εμπιστοσύνη των πολιτών της Μοσούλης και αυτό είναι σημαντικό διότι οι θρησκευτικές πολιτικές της χώρας και η έλλειψη εμπιστοσύνης στην περιοχή ε, επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2014 να μπορέσει να καταλάβει την περιοχή ο ISIS. Ε, αν καταφέρουν να παράσχουν κράτος ε, δικαίου και σωστή διακυβέρνηση και να δημιουργήσουν θεσμούς όπως ε, πανεπιστήμια. Δεύτερον, τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δωρήτριες χώρες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ταμείο για τη σταθεροποίηση και την οικοδόμηση της Μοσούλης η ε, ανθρωπιστική βοήθεια και οι ανάγκες ε, ανοικοδόμησης είναι τεράστιες και όλες αυτές οι χώρες μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο δεσμευόμενες να παράσχουν τα απαραίτητα ε, οικονομικά μέσα ούτω ώστε να δείξουν ότι δεν θα μείνει μόνη της η Μουσούλη. Τρίτον, οι ε, περιφερειακές και οι διεθνείς δυνάμεις θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ένωση παρά στην ε, ε, ένταση των διαφορών και θα πρέπει να οθήσουν την διανομή εξουσία στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χασάν. Μόλις μας ενημέρωσαν πως ο κύριος Ντεπράουερ χρειάστηκε να συμμετάσχει σε μια επίγουσα συνάντηση, οπότε δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα. Έχουμε εδώ εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα μου έχουν πει πως έχουμε εδώ τον επικεφαλής της ομάδας από ε, την ε, Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Έχουμε τον κύριο Γιώπης Φαν Κίρσμαν, ο οποίος ενδεχομένως θέλει να πάρει το λόγο και να μας πει ποια είναι τα αναπτυξιακά θέματα που προκύπτουν. Λέγομαι Φων Κίρχαμαν και είμαι ο τμήματάρχης ε, υπεύθυνο για θέματα Κεντρικής Ασίας, Μέσης Ανατολής, Κόλπο και Ειρηνικό και νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή που γίνεται. Να σας ευχαριστήσω και για τα όσα είπατε. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράσατε και πρέπει να σας πω και ως Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ε, φοβόμαστε πως η ήττα του ISIS στη Μοσούλη δεν αποτελεί και το τέλος αυτής της ιστορίας και, ιστορίας και αυτή η συμμαχία που μάχεται τον ISIS μπορεί ενδεχομένως να διασπαστεί και να οδηγήσει σε νέα προβλήματα στο μέλλον. Τώρα, για το δεύτερο σημείο που είπατε, πάνω σε αυτό, δηλαδή στο ότι οι δωρητές θα πρέπει να δημιουργήσουν ενδεχομένως ένα ειδικό ταμείο που θα έχει τα μέσα για να βοηθήσει, θα ήθελα πάνω σε αυτό να κάνω κάποια σχόλια. Σας υπενθυμίζω πως το Ιράκ ακόμα θεωρείται κράτος μέσω ανώτερου εισοδήματο. Οπότε για αναπτυξιακή βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη η επιλεξιμότητά του. Και αυτό έγινε το 2012 και 2013, όπου η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που ισχύει σήμερα. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν το Ιράκ σε τροχιά ελπιδοφόρα, τροχιά προς τη σταθερότητα και ήταν και οι τιμές πετρελαίου 118 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα είναι 34, οπότε καταλαβαίνετε πως αυτά είναι πολύ διαφορετικά. Και τα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας είναι πολύ περιορισμένα. Πριν σας πω ποια είναι τα σχέδιά μας, Θέλω να σου πω πως ελπίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να λάβει τα κονδύλια που είναι απαραίτητα του Ιράκ, τα οποία θεωρούμε εμείς πως είναι απαραίτητα μετά την ανακατάληψη της Μοσούλης για να σταθεροποιηθεί το Ιράκ. Να σας πω ποια θα είναι η δική μας παρέμβαση. Μ, αναφερθήκατε πως είμαι στην ΤΕΦΚΟ, αλλά πρέπει να σας πω πως για την περίπτωση του Ιράκ συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία Εξαιρετικής Εξωτερικής Δράσης, με την ΕΚΟ και με άλλες υπηρεσίες και ελπίζω στο μέλλον και με τα κράτη-μέλη, τα οποία είναι δραστήρια στην περιοχή του Ιράκ και νομίζω ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε κάτι το οποίο εμείς θα χαρακτηρίσουμε ως σφαιρικό σχέδιο δράσης για τη μετά Μουσούλη εποχή και δεν περιορίζεται στη Μοσούλη, αλλά θέλει να σταθεροποιήσει ολόκληρο το Ιράκ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε ποια είναι η σωστή αλληλουχία βημάτων και ελπίζω ότι σε μερικούς μήνες θα είμαστε σε θέση να έχουμε απόλυτη πρόσβαση στη Μοσούλη που θα είναι πάρα πολλές οι ανθρωπιστικές οι ανάγκες. Κρίμα που δεν είναι εδώ ο Ζαν Λουί γιατί πιστεύω πως η ΕΚΟ θα είναι ε, ο βασικός μοχλός ε, που θα κινήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Μοσούλη. Τούτου λεχθέντος πιστεύω πως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ε, στείνοντας ε, το όλο οικοδόμημα για μια μια μακροπρόθεσμη παρέμβαση και πιστεύω πως ένα βήμα που θα είναι απαραίτητο για να σταθεροποιηθεί το Ιράκ είναι να βασιστούμε στην ανθρωπιστική δράση που αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή η ΕΚΟ και μετά ένα τρίτο βήμα όπου εμείς πιστεύουμε πως θα πρέπει να βοηθήσουμε το Ιράκ να χρησιμοποιήσει τους δικούς του πόρους. Ας μην ξεχνάμε, το Ιράκ είναι μια χώρα πλούσια σε πόρους. Οπότε οι προσπάθειές μας μακροπρόθεσμα θα έπρεπε να είναι να βοηθήσουμε το Ιράκ να χρησιμοποιήσει αυτά που έχει στη διάθεσή του και να γίνει πάλι πολύ σταθερό. Παρόλο που ενδεχομένως αυτό είναι κάτι για το μακρινό, απότερο μέλλον. Βέβαια, είναι πολύ καλός υποψήφιος το Ιράκ για μέσα όπως το blending για την ανθρωπιστική βοήθεια, όπου χρησιμοποιούμε τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουμε για την προσπάθεια ανοικοδόμησης μιας χώρας γιατί υπάρχουν, επαναλαμβάνω, οι πόροι στο Ιράκ. Το σχέδιό μας λοιπόν θα περιγράψει τις διάφορες φάσεις και μετά θα προσπαθήσει να κάνει πιο συμπληρωματικές τις δράσεις όλων των υπηρεσιών μας με τον πιο πλήρη τρόπο. Θα κλείσω εδώ και όπως είπα και προηγουμένως ήρθα σήμερα και εγώ για να με στηρίξει το Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσετε να βρούμε διαθέσιμα κονδύλια για το Ιράκ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση σας αυτή. Θα ήθελα και πάλι να με συγχωρέσετε που δεν ε, μπόρεσα να προφέρω σωστά το όνομά σας. Ε, δεν είχα ενημερωθεί και ε, στην ώρα μου για το τι θα είστε παρόν. Τώρα έχουμε και εκπρόσωπο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης εδώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω στα πολύ γρήγορα και θα απηχήσω τα όσα είπε ο συνάδελφος κ. Φορκίρ Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η εκστρατεία για την Μοσούλη και τα όσα θα ακολουθήσουν δεν αποτελούν το, την αρχή του τέλους, απλώς το τέλος της αρχής και για τη διεθνή κοινότητα γιατί μετά τη Μοσούλη περίοδο θα πρέπει να μην αποστρέψουμε το βλέμμα μας από το Ιράκ όπως είχε γίνει μεταξύ του 11 και του 14 όπου είχαμε θεωρήσει πως ορίστε το Ιράκ είναι πλούσια χώρα ας βρει το δρόμο του ας ξεπεράσει μόνο του την αστάθεια, μεγάλο σφάλμα και ειδικότερα στο τρέχον, στην τρέχουσα συγκυρία, μια που έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη Συρία και οποιαδήποτε συνεχιζόμενη αστάθεια στο Ιράκ θα έχει επιπτώσεις και για τις γειτονικέ του χώρες. Οπότε πιστεύω πως όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα στη χώρα. Αυτή στο μέτρο του δυνατού. Για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Χασάν μίλησε για το Ταμείο για τη Σταθεροποίηση της Μοσούλης και αν υπάρχουν κονδύλια, γιατί εμείς έχουμε κάποια μέσα χρηματοδότησης για τη σταθεροποίηση, ας τα χρησιμοποιήσει. Το πρόβλημα είναι η ανασυγκρότηση, η ανοικοδόμηση, γιατί αυτή στο Ιράκ θα χρειαστεί πάρα πολλά δις και δεν είναι γνωστό από πού θα προέλθουν. Οπότε είναι μεν πλούσια χώρα το Ιράκ, ενδυνάμει πλούσια χώρα γιατί έχει πάρα, πολύ φυσικό πλούτο, αλλά ξέρετε πως οι μονάδες παραγωγής, πετρελοπαραγωγής, εάν δεν γίνουν ε, περαιτέρω επενδύσεις αυτή τη στιγμή ε, καταραίουν. Ξέρουμε πως οι πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να το κάνουν, αλλά με την τιμή πετρελαίου εκεί που είναι σήμερα δεν νομίζω πως η αγορά αυτή τη στιγμή τρέχει ε, για να κλείσει δουλειές. Και βέβαια δεν θα καλύψει και όλες τις ανάγκες που έχει η κυβέρνηση για ανοικοδόμηση και επενδύσεις. Η ίδια η κυβέρνηση έχει περιορισμένες ε, δυνατότητες ε, επένδυσης γιατί έχει υπογράψει μέχρι το 2020 πρόγραμμα για δημοσιονομική εξυγίανση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οπότε είναι μια περίοδος λιτότητας για να το πω έτσι για το Ιράκ. Οπότε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο των επόμενων τριών ετών ποιος θα μπει στο παιχνίδι για να βοηθήσει τους Ιρακινούς. Νομίζω ότι πρέπει και να βοηθηθούν από μόνοι τους, δηλαδή να βοηθήσουμε εμείς το Ιράκ να ε, χειραγωγήσει τις δικές του δυνατότητες και να τις χρησιμοποιήσει, αλλά και εξωτερικής ε, στήριξης, όχι απαραίτητα μέσω χρηματικών κονδυλίων, αλλά ενδεχομένως λύσεις για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του Ιράκ βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα βεβαίως είναι άλλες οι προοπτικές. Κλείνω εδώ. Thank you for your... Σας ευχαριστούμε. κύριος Στετίνα είναι ο πρώτος ομιλητής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ναι, ναι, βρείτε τα ακουστικά σας για να μιλήσω τη γλώσσα μου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χασάν. Κυρίως ε, για την παρουσίαση που μας κάνατε. σε σχέση με την ε, μεταμοσούλ εποχή, μετά την πτώση Μοσούλης. Ετέθη και το ζήτημα πόσο μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε το Ιράκ. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι η χώρα μου, η Τσεχική Δημοκρατία, πέρσι και πρόπεση. έδωσε στους Πεσμέργα 500 τόνους προμαχικά. Λίγαν ευκαταφρόνητη η υποστήριξη για την ε, ανακτήση της Μοσούλης. Δύο ερωτήσεις προς εσάς. Στον ε, αγώνα ε, για τη Μοσούλη ε, επεμβαίνουν και κουρδικές μειονότητες. Οι Σύριοι οι Κούρδοι είναι σίγουρα εκεί πέρα. Άλλοι Κούρδοι. Και δεύτερη ερώτηση, ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Έχουμε ακούσει πως ο τουρκικός στρατός είναι ε, στη Συρία, στα δυτικά του Εφράτη. Τι γίνεται με το βόρειο Ιράκ. Δεν μιλάω τώρα για το βομβαρδισμό των καταβλισμών ε, του ΠΚΚ. Ε, αυτή είναι παλιά ιστορία. Εγώ εννοώ αν συμμετέχει ο τελικό στρατό στην προσπάθεια απελευθέρωση Μοσούλη. Ευχαριστούμε. Καν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χάσαν που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας. Ε, και εγώ ερωτήσεις έχω για την μετά ε, την ε, ε νίκη κατά του ΑΣΥΣ. Ε, Μιλήσατε κυρίως για θέματα εμπιστοσύνης και καλής διακυβέρνησης στη Μουσούλη. Ξέρουμε από την ιστορική εμπειρία πως ε, ε, χρησιμοποιείται ε, οποιαδήποτε αποτυχία ε, ως γόνιμο έδαφος ε, για να ριζώσει περαιτέρω ο ISIS στην περιοχή. Ελαμβάνετε εσείς μέτρα για να μην επαναληφθεί δυστυχώς η ιστορία και πάλι. Και ένα συναφές ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, πόσο αποτελεσματική. Είναι η πρόσφατη ανακοίνηση σε σχέση με τις μάχημες ε, ομάδες ε, ΣΥΤΟΝ ε, που τελικά τώρα λειτουργούν υπό την αιγύδα του Πρωθυπουργού. Ε, κατά πόσο πιθανό θα ιτηθεί ο Αλτέζ. Και δύο είναι τα ζητήματα λοιπόν. Τι είναι με τον κατακαιρματισμό του Αλτέζ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις. Γιατί έχουν, από ό,τι ξέρουμε, και χημικά όπλα και ε, ακόμη χειρότερο την ικανότητα παρασκευής αυτών. Θέλω κι εγώ να απηχώντας την ερώτηση του κυρίου Χάν να επανέλθω ε, στη σύγκρουση στη Μοσούλη. Η επίθεση γίνεται από τρεις πλευρές ταυτόχρονα. Στα πρώτα στάδια της μάχης με ιδιαίτερες δυσκολίες κατελήθησαν αυτά τα χωριά με πολλά θύματα. Η μάχη σε αστικό περιβάλλον φυσικά είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έχετε στοιχεία για τα θύματα? Οι Ρακινές αρχές έκαναν Ανακοινώσει ε, θετικές και είπαν ότι νωρίτερα από το προσδοκόμενο σημειώθηκε επιτυχία, ξέρουμε. Τώρα όμω πως η σύραξη θα είναι παρατεταμένη και θα ισχύσουν ε, και διαφορετικοί όροι γιατί αλλάζει ο ρόλος του Αλτέζου. Μετά την εξαπόλυση της επίθεσης κυκλοφόρησαν φήμες πως ο ηγέτης ε, ε, έχει φύγει από την πόλη και έχει πάει ε, στην έρημο αφήνοντας τους λογαπού μαχητές που είναι προσιλωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Τι μπορείτε να μας πείτε για την ίδια τη μάχη Μετά την κατάληψη της Μοσούλης θα πρέπει να προγραμματίσουμε δραστηριότητες ανοικοδόμησης, αποκατάστασης εδαφών. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ξαναρχίσουν τη ζωή τους εκεί. Επίσης, αυτή η φέρπουσα υποψία ότι θα ενδεχομένω να χρησιμοποιηθούν όπλα μαζικής καταστροφής. Ε, πώς θα σχολιάζατε αυτό το, αυτή την υποψία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Χάσεν για αυτά που μας περιέγραψε. Αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει το οικονομική διάσταση ε, του ζητήματος προς τον ΑΛΤΑΕΣ. Υπάρχουν περίπλοκες αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικές μέθοδοι χρηματοδότησης ε, του ΝΤΑΕΣ από ό,τι έχουμε μάθει. Η αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης του ΝΤΑΕΣ Ε, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως βάση για να προβλέψουμε την μελλοντική ε, λειτουργία του ΝΤΑΕΣ, κυρίως ως προς την απόκτηση επιπρόσθετων στρατιωτικών ικανοτήτων. Οι χρηματοδοτικές πηγές είναι η πώληση πετρελαίου, δωρεές από άλλα κράτη, Έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στην οικονομική κατάσταση του ΝΤΑΕΣ. Κύριε Φασάν. Εδώ, εδώ είμαι. Στα δεξιά σας. Στα αριστερά σας μάλλον. Έχω δύο απλές ερωτήσεις. συναφής. Ε, στην αρχή της επίθεσης προβλέψαμε μαζική εκροή προσφύγων από τη Μοσούλη λόγω των ε, συγκρούσεων. Δεν ακούσα τίποτα σχετικό. Στην παρουσίασή σας έχετε στοιχεία για τους εκτοπιστέντες. Δεύτερον. Τι κάνατε για να αποτρέψετε την εισβολή στους καταβλισμούς προσφύγων των ξένων μαχητών. Γιατί έτσι εγκαταλείπουν και φεύγουν από τη Μοσούλη χωρίς, ε, χωρίς ποτέ να τιμωρηθούν για αυτά που έχουν κάνει. Ευχαριστούμε. Λόχ Μπίλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, ΕΚΟ, παρότι δεν εκπροσωπείται εδώ, διότι διευκόλυνε την επίσκεψη της υποφαινομένης και της βοηθού μου στην ε, Μοσούλη τον Οκτώβρη και σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε την ΕΚΟ διότι μας έδωσε ε, έγκυρα στοιχεία και ε, επιμελητιακή υποστήριξη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χασάν και άλλους ε, για την Τάλαφα. Κεντρωθήκατε στο ρόλο της πόλης και φαίνεται ότι ε, ο μόνο ο Ιρακινός στρατός λέει ότι χωρίς ε, τη, μια συγκεκριμένη μάχη, μια ομάδα που ήταν ιδιαίτερη αβάναυση μετά τη Φαλούτσα του Μάιο μπορούν να ε, καταλάβουν τη Μοσούλη. λένε ότι δεν θα ενταχθούν στο στρατό, ε, αλλά θα παραμείνουν στην τάλαφα, ίσως για τους λόγους που προαναφέρατε. Εσείς έχετε ακούσει κάτι τέτοιο? Ε, στον ακούστηκαν επικρίσεις για σοβαρά εγκλήματα πολέμου κατά της ε, ε μάχημης ομάδας, ε, ε, παραστρατιωτικής ομάδας και υπήρχαν ε, παράνομες δολοφονίες στην μάχη της ε, ε από αυτούς τους ήτες. Για την εποχή με... Για την μετά τη Μοσούλη περίοδο Φαίνεται πως εκπρόσωποι της ε, κουρδικής ε, κυβέρνησης ε, είπαν πως ο πρόεδρος ζητά συμμετοχή στη διοίκηση, αλλά δεν σημειώνεται πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει. και προς την Επιτροπή και την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Από κάποια σουνητικά χωριά στο νότο Ε, μαθαίναμε ιστορίες ε, και τελικά τι γινόταν δύο χρόνια πριν. Ήταν εκτεθειμένα σε ακραία βία τα παιδιά εκεί τα σκοτώνουν και τα υποχρεώνουν να κάνουν πράγματα που δεν αρμόζουν σε παιδιά. Δηλαδή, ε, πρόκειται για σοβαρά τραύματα για ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Ε, οι διεθνεί οργανώσει με τι οποίε ε, συνομιλήσαμε είπαν ότι προετοιμάζονται για μεγαλύτερους αριθμού προσφύγων. Προς το παρόν τα καταφέρνουν. Έχουν δηλαδή θεραπεία για μετατραυματικέ ε, εμπειρίε. Τώρα που έχει κατάσταση. Τότε μας είπανε δεν έχει νόημα να πάτε στις Βρυξέλλες για να ζητήσετε ε, χρηματοδότηση. Γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσοι θα είναι οι πρόσφυγες ε, προς το παρόν. Σας ευχαριστούμε. Κύριε αν μπορείτε να απαντήσετε... Ε, στις ερωτήσεις των ε, βουλευτών. Κυρία Κίσμαν. Και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, αν προτίθεται να απαντήσει τι ερωτήσεις, θα σα δώσω το λόγο αμέσω μετά. Ο κύριο Καβαχασάκη. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Θα ξεκινήσω ε, σχετικά ε, με τις παρεμβάσεις των κυρίων από την ΕΦΚΟ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Συμφωνώ απόλυτα ότι το ε, Ιράκ είναι ε, μια χώρα με πόρους, ε, όχι μόνο πετρέλαιο αλλά και ανθρώπινους πόρους. Έχει περήφανο λαό, μεγάλο πολιτισμό, όλα αυτά ισχύουν. Όμως ταυτόχρονα η πικρή αλήθεια είναι ότι το Ιράκ βρίσκεται ένα βήμα πριν της χρεοκοπίας και αυτό ε, έρχεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που έχει τη μάχη κατά του ISIS, όμως βέβαια τα πηγαίνει κάπως καλύτερα σε σχέση με το Κουρδιστάν. Ας φανταστούμε λοιπόν σε έξι μήνες ε, ε, η Μουσούλη θα έχει απελευθερωθεί, ο Άισις θα έχει ιτηθεί. Η Ιρακινή κυβέρνηση ως γνωρίζουμε δεν έχει τους οικονομικούς πόρους για να μπορέσει να ε, κάνει τα έργα τα οποία χρειάζονται άμεσα για την σταθεροποίηση στην Μουσούλη. Δεν υπάρχουν τα χρήματα και έτσι λοιπόν θα υπάρχει μεγάλη διαφθορά όπως είπες και στο Κρατζή Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτό το οποίο χρειάζεται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ε, να υπάρχει ε, χρηματοδότηση με βάση όρους που θα βασίζεται δηλαδή στο κράτος δικαίου, δικαίου την, καλή, την διακυβέρνηση, τη μετάβαση εξουσίας την αποτροπή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει, ο καθένας θα πρέπει να διώκεται, κανένας δεν είναι υπεράνω νόμου και δημοσίως θα πρέπει να φανεί στους πολίτες ε, της χώρας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα για να βοηθήσει. Και η κυβέρνηση βέβαια έχει την ευθύνη. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καμία άλλη εναλλακτική πέραν αυτής, τουλάχιστον ε, χρηματο, ε, χρηματοδοτική υποστήριξη για 2-3 χρόνια με βάση αυτά τα γενικά κριτήρια στον κύριο Στρέτσινα. Ευελπιστώ να έχω προφέρει σωστά το όνομά σας. Οι ε, Κούρδοι αγωνιστές από τη Συρία, τη Ροζάβα, συμμετέχουν στις μάχες, όχι το ΠΚΚ. Όπως ε, γνωρίζουμε βρίσκεται σε περιοχές του ε, δεν έχουν συμμετάσχει ακόμα στη μάχη της Μουσούλης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, διεξάγουν ένα πάρα πολύ καλό συντονισμό μεταξύ όλων αυτών των ε, παρατάξεων με αποτέλεσμα να μειωθούν οι εντάσεις ε, για την ώρα. Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν ε, εντάσεις μεταξύ του ΚΑΔΕΠΕ και του ΠΚΚ και γι' αυτό το λόγο τους ε, κρατούσαν τις παρατάξεις χωρισμένες, όμως αυτό έχει επιληθεί για την ώρα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν συμμετάσχει στη μάχη της Μοσούλης ε, αυτή καθ' αυτή. Τώρα αν υπάρχει επιρροή από την πλευρά της Τουρκίας, ναι, σίγουρα όπως γνωρίζουμε ναι, τα στρατεύματα, τα στρατεύματα που έχουν στο Βασίλειο δεν είναι τόσο μεγάλα, 3-4 χιλιάδες ε, στρατιώτες, ε, όμως ε, τα μηνύματα, τα πολιτικά μηνύματα από την πλευρά της Άγκυρας, αλλά και την πιθανότητα μίας διαμάχης με το Ιράκ θα πρέπει να τονίσουμε ότι στρατεύματα της ΙΑ θα καταλάβουν το Ταλάφαρ και τότε να περιμένουμε περισσότερη παρέμβαση από την πλευρά της Τουρκίας και ε, θα υπάρχουν συνέπειες τόσο για το Ιράκ όσο βέβαια και για την Τουρκία αλλά και για άλλες χώρες της περιοχής. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη, ε, κύριε Χάν, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και βέβαια είναι δύσκολο ε, να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη όταν έχει χαθεί. Ισχύει για τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και ισχύει και για τη σχέση μεταξύ ε, πολιτείας και κοινωνίας. Ε, οι Ρουάχοι γενικότερα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν, ζουν σε ειρηνικές περιοχές έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους ε, παρόλο που έχουμε εκλογές ε, στο Ιράκ ε, υπάρχει αυτή η δυσλειτουργική δημοκρατία στη χώρα και παρόλο που υπάρχουν ισχυρισμοί για ζητήματα διαφθοράς και όταν μιλάω για διαφθορά δεν εννοώ μικροδιαφθορές αλλά σε, όλο το φάσμα της πολιτικής ελίτ που παρουσιάζεται μετά το 2003 μπορεί να ανοικοδομηθεί και πάλι. Νομίζω ότι βλέπουμε κάποια πρώτα θετικά σημάδια από όλες τις πλευρές. Βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός Χαρμπάντη έχει την διάθεση ε, να στραφεί στους πολίτες ε, της Μοσούλης και τις διάφορες πλευρές. Είναι ειλικρινής για αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι επίσης υπάρχει συζήτηση για το ζήτημα του Ταλάφαρ έχουμε πιο μετριοπαθείς ομάδες ε, ΣΥΑ που θέλουν να συμμετάσχουν στη μάχη εάν ε, επιβληθούν εκεί ε, και αποτρέψουν ή εστοπίσουν τους, τις πιο σκληροπυρηνικές ομάδες τότε θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα όμως πάνω απ' όλα όσον αφορά ε, την επαναφορά της εμπιστοσύνης θα πρέπει να υπάρξει ε, ένα πραγματικό σχίσμα μεταξύ των πρακτικών διαφθοράς που υπήρχαν στο παρελθόν. Και παρά τα όλα, όλα τα δυσάρεστα νέα που μας έρχονται από το Ιράκ υπάρχουν και θετικές ιστορίες. Η κοινωνία των πολιτών γίνεται πιο ισχυρή καλούν ε, για κράτος δικαίου, ε, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές ε, και δυστυχώς αυτές οι φωνές δεν εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς. Όταν έχουμε τις μάχες σχετικά με το Μοσούλη υπάρχουν μονάχα τα αρνητικά νέα τα οποία επικεντρώνονται στην, ε, στην όλη διήγηση. Δεν είναι χαμένη υπόθεση λοιπόν, ε, υπάρχει δυνατότητα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της χώρας ε, για να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Και σας μιλάω τώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που υπάρχει ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο και στρατηγική για την υποστήριξη του Ιράκ που θα βασίζεται σε συγκεκριμένους όρους όπως είναι για παράδειγμα το κράτος δικαίου. Οι νόμοι που ε, περάστηκαν στο Κοινοβούλιο αφορούν την υπεράσπιση της ε, κοινωνίας. Οι Σουνίτες δεν συμμετείχαν ε, στην ψηφοφορία. Οι Κούρδοι, περισσότεροι εξ αυτών το υποστήριξαν και χθες προχθές ε, ο Πρωθυπουργός Μπαρζάνη είπε ότι χαιρετίζουν το συγκεκριμένο νόμο όμως ας δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά και ποια θα είναι η επιρροή τους ε, στη σχέση μεταξύ των Σουνιτών και των ΣΥΑ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ε, νωρίς ε, για να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες του συγκεκριμένου νόμου. Όσον αφορά τα όπλα μαζική καταστροφής, ναι, όντω αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ε, κίνδυνο και όπως φαίνεται από αναφορές του Άσις φαίνεται ότι έχουν ε, την ικανότητα και το έχουν ε, δείξει σε διάφορες τοποθεσίε στο Ιράκ, τόσο εναντίον αμάχων όσο και στρατευμάτων. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, όμως ε, και με βάση τις επαφές μου στο Ιράκ, ε, αλλά και ε, διάφορους άλλους επαγγελματίες διεθνώς, Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις ικανότητες του ISIS, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό, όμως παραμένει μια μεγάλη ε, απειλή τόσο για τα στρατεύματα όσο και για τους αμάχους. Για ποιο λόγο δεν μίλησε για τους πρόσφυγες, καλό ερώτημα, διότι ζητήθηκα να επικεντρωθώ στην πολιτική και στρατιωτική διάσταση της ε, διαμάχης ε, και πιστεύω ότι ο κύριος Ντεπράουρ ζητήθηκε να επικεντρωθεί στην ανθρωπιστική διάσταση της διαμάχης και όσον αφορά την προσφυγική κρίση και γι' αυτό το λόγο δεν επικεντρώθηκα στο ζήτημα των προσφύγων. τα ε, τραυματισμένα παιδιά δεν είναι μονάχα παιδιά, τα παιδιά που έχουν, φέρουν ένα τραύμα, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία και τα παιδιά και οι ενήλικες. Και νομίζω ότι τα επερχόμενα χρόνια, ίσως και δεκαετίες, εκτός από την ανοικοδόμηση, το κράτος δικαίου, θα χρειαστεί και ένας ολόκληρος στρατός ψυχολόγων, θεραπευτών για να βοηθήσουν τους Ιρακινούς ε, να ανταπεξέλθουν ε, με όλα αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί από τον ISIS και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι κομμάτι της όλης προσέγγισης ε, σχετικά με το Ιράκ μετά την απελευθέρωση της Μοσούλης. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι ενός σχεδίου όχι μονάχα για την ανοικοδόμηση δρόμων, σχολείων, αλλά και την ανοικοδόμηση της προσωπικότητας του Ιράκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Ντεμπράουρ από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ξέρω πως ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και για εμένα. γιατί εγώ ήρθα από τον Κτάσκο που είχαμε χιονωθεί, αλλά και όπου ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις, οπότε και εγώ καθυστέρησα με τη σειρά μου. Ελπίζω όμως πως θα καταφέρουμε να φτάσουμε επιτυχώς μέχρι το τέλος της σημερινής ε, συνειδρίασης, γιατί είναι σημαντικά τα συμπεράσματα στα οποία θα στα οποία θα καταλήξουμε. Θα ήθελα να καλέσω και τον κύριο Χάρισον και τον κύριο Κίρχμα να σχολιάσουν και μετά θα δώσω το λόγο στο διευθυντή κύριο Ντεμπράουερ για να μας πει δύο λόγια. Για ερωτήσεις μετά θα έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά έχουν ήδη έρθει οι ομιλητές για το επόμενο θέμα και δεν θα ήθελα να τους καθυστερήσω υπερβολικά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας και μπορώ να σας απαντήσω ήδη πως τέτοιου είδους ε, παρεμβάσεις για παιδιά τα οποία έχουν τραυματικές εμπειρίες είναι κομμάτι αυτών που κάνουμε στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδίου και φυσικά κάτι τέτοιο αποτελεί κομμάτι για το κατά πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί δίνοντας περισσότερα χρήματα στο Ιράκ. Αυτό κατάλαβα ότι είπατε. Ναι, Κοιτάξτε, τα χρήματα τα οποία επενδύουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια και τα οποία θα φτάσουν δύο, μετά από δύο-τρία χρόνια στην οικονομία, ελπίζω πως θα επιτρέψουν στο Ιράκ να ξαναγυρίσει σε τροχιά σταθερότητας. Και γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η ενδιάμεση παρέμβαση, αλλά καλό είναι να υπάρξει και βοήθεια άμεση έτσι ώστε ε, μακροπρόθεσμα να είναι αυτόνομο σε αυτό το επίπεδο το Ιράκ. Τώρα για την ε, υποπροϋποθέση στήριξη, να σας πω, όταν η στήριξη βασίζεται για παράδειγμα στην απόδειξη της χρηστής διαχείρισης από μια κυβέρνηση, κοιτάξτε, για άμεση παρέμβαση αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγάλες ανάγκες, και ο κύριος Ντεμπράουερ θα μας τα πει αυτά, Είναι δύσκολο. Πάντως για τα μέσο μακροπρόθεσμα αυτό ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή μία παρέμβαση στο Ιράκ που θα σχετίζεται και θα συνδέεται με αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε δείκτες και ένας από αυτούς τους δείκτες συνήθως είναι και η καλή διακυβέρνηση. Και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Το Ιράκ είναι σε πολιτιστικό επίπεδο εξαιρετικά πλούσια χώρα αλλά δεν είμαι σίγουροι πως είναι τόσο πλούσια σε ανθρώπινους πόρους. Εγώ ήμουνα τέσσερα χρόνια στο Ιράκ και πρέπει να σας πω πως ήδη εκείνη την εποχή είχαν τεράστια διαρροή εγκεφάλων. Δεν νομίζω σήμερα πως θα έλεγα πως έχουν τόσο πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό. Ελπίζω όμως πως το μέλλον θα επιστρέψουν. Σας ευχαριστώ. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα πω πως για την αιρεσιμότητα, δηλαδή την υποπροϋποθέση στήριξη για την ανθρωπιστική βοήθεια αυτή δεν μπορεί να βασίζεται σε προϋποθέσεις. Πάντα είναι χωρίς προϋποθέσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Θα το πει και ο διευθυντή μας και για την στήριξη σταθερότητας όχι μόνο από την ΤΕΦΚΟ αλλά και από άλλους πρέπει να σου πω ότι συνδέεται τόσο πολύ με τις άμεσες ανάγκες που χρειάζεται να στηρίξουμε ανεξάρτητα με το πώς πάνε τα πράγματα στο Ιράκ. Να σας διαβεβαιώσω πως όποτε γίνονται συζητήσεις με τις Ιρακινές αρχές για τη σταθεροποίηση είτε για κάποιο άλλο θέμα, για το κράτος δικαίου, για τις δυνάμεις ασφαλείας, πάντα μιλάμε για το θέμα της διακυβέρνησης, ορθής διακυβέρνησης. Είναι το μάντρα που επαναλαμβάνουμε. Και αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί και τη γραμμή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεμπράουερ από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι πολύ που καθυστέρησα. Είχαμε αυτή τη στιγμή στρατηγικό διάλογο με τον Ερθρό Σταυρό όλη μέρα και ειδικά το θέμα του Ιράκ ήταν ψηλά στην ημέρη σε διάταξη, κυρίως για τις συνθήκες εργασίας. Με μεγάλη χαρά Είδα πως έχω εδώ συναδέλφους από την ΤΕΡΚΟ και από την Υπηρεσία Εξαιρετική Δράσης και ω εισαγωγή να σας πω πως ο τρόπος με τον οποίο εμείς τα όργανα στηρίζουμε την κατάσταση στο Ιράκ είναι μια πολύ καλή διαδικασία, συντονισμένη, αλληλένδετη και είναι πραγματικά εξαιρετικό το επίπεδο συνεργασίας που έχουμε επιτύχει. Και η κοινή μας παρουσία εδώ το αποδεικνύει. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω σε ποια απάντηση απαντούσατε όταν μπήκα. Πάντως αυτά που λέτε τα πιστεύω και εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν πιστεύω πως είναι χαμένη η υπόθεση στο Ιράκ. Όπως είπατε και εσείς. Δεν είναι. Και εμείς προσπαθούμε ως ανθρωπιστική διεύθυνση να το κάνουμε να επαληθευθεί, γιατί τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια έχουμε υπερασπιστεί την εξή σκέψη, πως θα πρέπει να είναι ουδέτερη, αμερόληπτη και κυρίως χωρίς προϋποθέσεις η ανθρωπιστική βοήθεια, να βοηθάει τους πιο ευάλωτους όπου να είναι, όποιοι και να είναι και με όποιο τρόπο γίνεται για οποιαδήποτε ανάγκη τους. Και δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ κοινοτήτων, μειονοτήτων ή άλλων. Είναι το κατά πόσο είναι ευάλωτη για να εξασφαλίσουμε πως σύμφωνα με το μάντρα της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Συνόδου και των στόχων να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Και αν υπάρχει μία χώρα στην οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν πίσω είναι το Ιράκ. Και θα πρέπει να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια με έναν τρόπο που θα συνεισφέρει έτσι ώστε να μείνει κάποιο είδους κοινωνικός ιστός σε μια χώρα έτσι ώστε να επανακάμψει στο μέλλον. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα όσα οργάνωσε σήμερα το απόγευμα και είστε κι εσείς δημοσιονομική αρχή και σας ευχαριστώ για τη γενοδορία σας γιατί κάνατε μια θετική αξιολόγηση του αιτήματο για τροποποιητικό προπολογισμό και έτσι θα μπορέσουμε στο Ιράκ και κοντά στη Μοσούλη να αυξήσουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια πριν τα τέλη του έτους. Για την ίδια τη Μοσούλη, όπως ξέρετε κι εσείς, το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι πως το βλέπαμε. Το βλέπαμε να γίνεται και είχαμε σχέδια έκτακτης ανάγκης τους τελευταίους έξι μήνες. Για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της μάχης της Μοσούλης είχε σκοπό να ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου και όντως 17 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι πως το μόνο σενάριο στο οποίο είχαμε οικοδομήσει αυτό είναι τεράστιες ροές να εγκαταλείπουν την πόλη και αυτό δεν έγινε. Γιατί? Γιατί και οι Ρακινές δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις που το στηρίζουν έχουν ακολουθήσει μια τακτική επιχειρήσεων πολύ ενδιαφέρουσα με ένα τελείως διαφορετικό σενάριο προστασίας, προστασία μάχων εκεί που βρίσκονται, χωρίς να ε, υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Και μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που το μέτωπο έφτασε τα προάστρια της Μοσούλης, ήταν έτσι. Οπότε ήταν περιορισμένος μάλλον ο αριθμός των εκτοπισμένων, όταν λέω περιορισμένος, είναι περίπου 70.000 άνθρωποι, αλλά πολύ χαμηλότερο αυτό το νούμερο από τις αρχικές μας προβλέψεις. Τούτου λεχθέντος πήγα στην χωράγια κοντά στη Μοσούλη πριν από τέσσερις εβδομάδες και το είπα ανοιχτά και το ξέρουν οι εταίροι μας θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει καλύτερη ανθρωπιστική απόκριση. Παρόλο που έχουμε αυτά τα σχέδια έκτακτη ανάγκης, γιατί είχαμε πολλά κενά. Και με χαρά βλέπω πω οι περισσότεροι εταίροι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν κάποια αυστηρότητα στον προγραμματισμό τους, γιατί είχε ως σκοπό η ανθρωπιστική βοήθεια να καλύψει μεγάλους όγκους πληθυσμού και όχι μια κατάσταση όπου ελάμβανε χώρα σε χωριά, σε πόλεις που απελευθερωνόταν το ένα μετά το άλλο από τις Ιρακινές δυνάμεις. Οπότε ήταν μια μάλλον δύσκολη στιγμή για την ανθρωπιστική κοινότητα, όμως ευτυχώς τα πράγματα βελτιώθηκαν και πάνε καλύτερα. Είμαστε πάλι στο σωστό δρόμο και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει στο να αποκριθούμε στις ανάγκες, ακόμα κάποια κενά πρέπει να καλυφθούν κλάδους υγείας, τραυματίες, ε, άνθρωποι με τραυματικές εμπειρίες, αλλά το συζητάμε με τον Ερυθρό Σταυρό, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα και τους έχουμε ζητήσει να επανεπενδύσουν στην γειτονιά αυτή έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και αυτές τις ανάγκες. Μέχρι σήμερα αυτό που είδαμε είναι πως πρόκειται για πόλεμο. Δηλαδή είναι ένας πόλεμος αλλά οι Ιρακινές δυνάμεις και οι ένοπλες ομάδες και οι κουρδικές ένοπλες ε, ομάδες έχουν σεβαστεί αυτά τα οποία είχαν ε, συμφωνήσει. Τώρα, έχουμε πρόβλημα με τη διαδικασία screening. Έχουμε αμφιβολίες γιατί για τους ίδιους ήταν βασικό να μπορούν να κάνουν ένα screening για να ξεχωρίσουν αυτούς που εγκαταλείπουν τη Μοσούλη για να είναι σίγουροι πως από αυτούς που εγκαταλείπουν δεν ήταν μαχητές. Οπότε είχαν συμφωνήσει ένα διάφανο, μια διάφανη διαδικασία screening, το οποίο εντάξει χρειάστηκε χρόνο, έτσι για να το πω ευγενικά. Αυτό που ακούω από τον Ερυθρό Σταυρό σήμερα, ότι και στη Μοσούλη και στην περιοχή γύρω από τη Μοσούλη, είναι πως αυτή η διαδικασία screening έχει στηθεί, εφαρμόζεται με σχετικά διάφανο τρόπο, αλλά αυτό το οποίο ακόμα δεν είναι όπως θα έπρεπε είναι οι συνθήκες κράτησης για αυτούς οι οποίοι έχουν αποτύχει στο screening, δηλαδή έχουν ταυτοποιηθεί ως μαχητές. Όπου ο Ερυθρός Σταυρός έχει καταρχήν πρόσβαση σε κάθε εγκατάσταση κέντρο κράτησης, αλλά ακόμα αυτό δεν έχει εφαρμοστεί. Τώρα, τι οψή έχει το μέλλον. Και μου είπατε να είμαι σύντομος, θα το πω τηλεγραφικά. Μπαίνουμε τώρα σε μια διαφορετική φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η πόλη έχει σχεδόν ε, περικυκλωθεί και έχουν ξεκινήσει οι μάχες μέσα στο ίδιο το αστικό περιβάλλον. Καταστράφηκαν οι πρώτες γέφυρες πάνω από τον ποταμό και είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα για όλους και πολύ πιο επικίνδυνο για τους αμάχους. Οπότε μπορεί να αλλάξει η αρχή της επιχείρησης και αντί να προσπαθήσουν να κρατήσουν τους ε, ε, κατοίκους εκεί που βρίσκονται και να τους προστατεύσουν εκεί, μπορεί να περάσουμε σε ένα σκεπτικό που είναι σαν τα όσα είχαμε στη Φαλούτζα, δηλαδή θα κληθούν όλοι να εγκαταλείψουν μαζικά την πόλη πριν να βομβαρδιστεί μέχρι να γίνουν όλα συντρίμια από τις Ιρακινές δυνάμεις και βέβαια και από τις ενοπλές ομάδες. Αυτό θα φανεί. Έχουμε αυτές τις φήμες που κυκλοφορούν, αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα επίπεδα βίας εντατικοποιούνται εντυπωσιακά και βέβαια οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν λάβει τελείως διαφορετική μορφή, μια και λαμβάνουν χώρα μέσα στην ίδια την πόλη. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε στενά, γιατί πολύ άσχημες οι αναμνήσεις από το Ραμάντι και τη Φαλούτζα και κανείς δεν θα ήθελε αυτό να ξανασυμβεί. Θα παρακολουθήσουμε στενά λοιπόν τις εξελίξεις εμείς στη διεθνή κοινότητα. Τώρα, ο νόμος που πέρασε για τις ένοπλες δυνάμεις χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο, καθυστέρησε. Είναι επιτυχία το ότι ψηφίστηκε. Αυτές οι ένοπλες δυνάμεις λένε πώς θα ακολουθήσουν τα όσα του ζήτησε ο Πρωθυπουργό. Θα μείνουν σε δεύτερο, ε, σε δεύτερο ρόλο και δεν θα μπουν ούτε στη Μουσούλη ούτε στο Ταλάφα. Ελπίζω. Ελπίζω πως θα μείνουν έτσι λίγο πίσω και θα το κάνουν αυτό. Η εντύπωση μου είναι, συζητώντας μαζί τους, ότι αυτή είναι μια κατάσταση όπου όλοι έχουν το χέρι στη σκανδάλη. Οπότε και το μικρότερο επεισόδιο μπορεί τελικά να κλιμακωθεί σε έναν ανοιχτό πόλεμο. Ας είμαστε προσεκτικοί λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε υπερβολικά απεσιόδοξοι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος και μου Να παρακολουθούμε λοιπόν μέρα-μέρα το τι γίνεται. Τώρα, και ένα τελευταίο, ακολουθώντας τα όσα είπε ο συνάδελφος Φων Κίρσμαν, 16 Δεκεμβρίου θα γίνει μια συνάντηση στις Βρυξέλλες όπου θα έχουμε και ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις αλλά και εκπροσώπους της μεταβατικής ατζέντα, του μεταβατικού θεματολογίου γιατί βέβαια γίνεται μια τεράστια επένδυση στο μέλλον αυτής της χώρας και θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα ποια είναι τα σχέδιά μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα τα δύο μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να εργολοποιηθούν μαζί γιατί βέβαια η ανθρωπιστική βοήθεια θα χρειαστεί και για τη Μουσούλη και γύρω από τη Μοσούλη, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε με το που θα γίνει αυτό να προχωρήσουμε σε αποναρκοθετήσεις, ε, δημόσιες υπηρεσίες σε ένα ελάχιστο επίπεδο στην πόλη, γιατί έχουν καταστραφεί από τη μάχη που γίνεται και που θα συνεχίσει να γίνεται. Και επίσης ουσιαστικό είναι, επειδή έχει περικεκλωθεί η πόλη, να έχουμε κάποιες διόδους διαφυγής γιατί ωραία, να ζητήσουμε από τον πληθυσμό να εγκαταλείψει την πόλη και έτσι να μείνουν στην πόλη μόνο τα μαχόμενα μέρη, αλλά θα πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία να φύγουν. Και αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί. Και πρέπει να σα πω προς τις για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται εκεί καμία διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων που εγκαταλείπουν τη σύραξη και καταλαβαίνετε πως αυτό είναι ανησυχητικό για μας. για τα όσα θα συμβούν τις επόμενες εβδομάδες ή ημέρες. Σήμερα γίνονται επιθέσεις μέσα στη Μοσούλη, άρα λοιπόν ήταν πολύ επίκαιρη η σημερινή συζήτηση, γιατί όπως είπατε και εσείς, ακούσαμε διάφορα σενάρια. Ακολουθήσαμε άλλο σενάριο στην αρχή και τώρα νομίζω ότι έφτασε η στιγμή που θα περάσουμε σε μια άλλη φάση της μάχης, πιο δύσκολη, με πιο μεγάλες ε, επιπτώσεις για τα ανθρωπιστικά θέματα, για παράδειγμα σε πιο περίπλοκη πολύπλοκη πολιτική, πολιτική κατάσταση όταν θα έρθει η στιγμή ανοικοδόμηση της χώρας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεμπράουερ που καταρχήν ήρθατε και μιλήσατε. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν να ακούσουμε γιατί έκλεισε ε, τα... και βοήθησε την ενημέρωσή μας για το τι συμβαίνει στην πόλη αυτή και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση του Ιράκ. Και βέβαια όταν θυμάμαι τη συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως μετά την ε, κίνηση της επίθεσης στη Μοσούλη να σας πω πως πήραν το λόγο πάρα πολλοί ευρωβουλευτές και στήριξαν επιπλέον δημοσιονομική στήριξη μέσω του προϋπολογισμού. Εμείς αναγνωρίζουμε πως θα είναι μια μακρά διαδικασία και είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Φοβάμαι πως πρέπει να κλείσουμε στο σημείο αυτό της ημερής διάταξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν. Τον ε, κύριο Χασάν, τον κύριο Ντεμπράουερ, τον κύριο Φον Κίρσμαν, και τον κύριο Χάρισιον. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης αφορά την ενημέρωση σχετικά με την αποστολή ε, που κάναμε στην Ουκρανία μεταξύ της 1ης ε, και 4ης Νοεμβρίου και καθώς το συγκεκριμένο ε, θέμα σχετίζεται με το ε, επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης, την ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη Τζον Herbst, ο οποίος θα μιλήσει σχετικά με την κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία θα ήθελα να καλέσω τον ε, πρέσβη να έρθει να καθίσει εδώ μαζί μας ε, στο Προεδρείο, όχι ακριβώς στο Προεδρείο, όμως ε, θα ήθελα να τον καλέσω να καθίσει εδώ και να συζητήσουμε και για τα δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συνδυάσω τα επόμενα δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης ε, και θα ήθελα να καλέσω στην ε, συνεδρίασή μας ε, τον πρέσβη John Herbst, ο οποίος είναι Αμερικανός ε, διπλωμάτης που ε, τέλει ως πρέσβης ε, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ουσβεκιστάν και στην Ουκρανία. Ε, περιμένουμε λοιπόν τα σχόλια της εξοχότητάς του πάνω σε αυτά τα ζητήματα. τα οποία ε, μας απασχολούν τακτικά στις ε, συναντήσεις μας ε, τις Δευτέρες. Και το σημείο της ημερήσιας διάταξης το οποίο θα συζητήσει ο πρέσβης είναι η κατάσταση της ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία Τώρα ε, θα ήθελα να σας πω κάποια ε, πράγματα σχετικά με την πρόσφατη μας αποστολή στην Ουκρανία. Πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 1ης ε, και 4ης Νοεμβρίου. Συμμετείχαν τέσσερα μέλη της Υποεπιτροπής Ασφάλειας, καθώς επίσης ε, και διάφοροι πολιτικοί ε, σύμβουλοι και ε, μέλη της Γραμματείας. Ο κύριος Μάικλ Γκάλλερ συμμετείχε από την ΕΠΠ. Ο κύριος Βαν Μπάλεν από την Άλντε ο ε, καθηγητής ε, Μπούχνα από τους ε, Πράσινους και είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε την πολιτική, οικονομική, κοινωνική κατάσταση στην Ουκρανία καθώς επίσης και ζητήματα ασφαλείας ε, με ε, σημαντικούς ε, παράγοντες οι οποίοι εκπροσωπούν διάφορους τομείς της Ουκρανικής Αρχής. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο και τότε λοιπόν είχαμε την τύχη να ταξιδέψουμε και στα ανατολικά της χώρας κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι είχαμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε ε, προσωπικό από εκεί και να συζητήσουμε επίσης ε, με θύματα ε, μαχών στα ανατολικά της χώρας και στη συνέχεια πήγαμε στο Κράματόρσκ και ε, πήγαμε ακόμα πιο κοντά ε, στα παιδιά μάχης και εκεί μπορέσαμε να, να συζητήσουμε με διοικητές ε, στρατευμάτων, όπως επίσης και με ηγέτες της ομάδων κοινωνίας των πολιτών, με διάφορες ΜΚΟ που, που φροντίζουν τους ντόπιου πληθυσμούς και εκεί φυσικά είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια συζήτηση και ανταλλαγή από, ε, απόψεων με την αποστολή του ΑΟΣΑ στο Κραμαντόρσκ κάτι το οποίο επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρον. Επίσης μας δόθηκε η δυνατότητα να ε, επισκεφθούμε εγκαταστάσεις ε, υγείας ε, στην περιοχή που φροντίσουν τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Επίσης, η μία επίσκεψη επισκευ... ήταν επικεντρωμένη ε, στην ποιότητα παροχής υγείας ε, που ε, φροντίζει τόσο, για τους εσωτε... τόσο τους εσωτερικά εκτοπισμένους όσο και τους στρατιώτες και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν στις μάχες και βρίσκονται κοντά στο Ντονέτσκ ε, και το αεροδρόμιο του. Δεν ήταν μονάχα ενδιαφέρον, ε, αλλά ταυτόχρονα ε, λάβαμε πολλές πληροφορίες. Ο πρώτος γύρος συζητήσεων έλαβε χώρα στο Κίεβο και ξεκίνησε με ε, τις ε, ε, διπλωματικές εκπροσωπήσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθώς επίσης και με διπλωμάτες του ΟΑΣΑ και συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων, κυρίως όμως επικεντρωθήκαμε στο ζήτημα της ασφάλειας στην Ουκρανία, της, την, η Δευτέρα Νοεμβρίου ήταν αφιερωμένη ε, στην ε, πολιτική συζήτηση με τις αρχές της Ουκρανίας όπου συμμετείχαν ε, μέλη του Κοινοβουλίου και εκπροσώπους των Ταρτάρων ενώ την ε, δεύτερη φορά, ήταν η δεύτερη φορά που συναντήσαμε τον κύριο Τσαμάροφ, ήταν μια συνήθις ε, συζήτηση σχετικά με την κατάσταση ασφάλειας ε, όσον αφορά την ε, ε, Κρυμαία μετά την παράνομη προσάρτησή της και επικεντρωθήκαμε κυρίως ε, στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, κατά ε, συγκεκριμένων ομάδων της κοινωνίας καθώς επίσης και την κατάσταση για τους Τατάρους στην Κρυμαία. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει ένα ε, ψήφισμα αφιερωμένο στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή του Τατάρους της Κρυμαίας. Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά συναντήσεων όπως για παράδειγμα με τον επικεφαλή του τμήματος ε, ε, ε, Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Τούρτσινοφ, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι υπουργός υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τον, την κυρία Κλίμπους Τσιντσάτζε, όπως επίσης ε, και ε, τους επικεφαλείς ε, της Επιτροπής Ασφαλείας ενώ συναντήσαμε και τον Υφυπουργό Άνμινας και Εξωτερικών Υποθέσεων όλες αυτές οι συναντήσεις ήταν αφιερωμένος, αφιερωμένες στην κατάσταση ασφαλείας και τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ουκρανία. Η τελευταία συνάντηση ήταν με ένα άτομο το οποίο είναι αρκετά γνωστό σε εμάς. Είναι ε, αντιπρόεδρος ε, της ε, ε, προεδρικής Διοίκησης, ε, τον κύριο Κωνσταντίν Γελιέσιευ, κατά τη διάρκεια όλων ε, των συναντήσεων. Δύο ήταν τα ζητήματα τα οποία βρισκόταν στο προσκήνιο από την πλευρά της Ουκρανίας Το πρώτο λοιπόν ήταν ε, η απελευθέρωση των θεωρήσεων και η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ξεκάθαρη πάνω σε αυτό. Εμείς οι τέσσερις εκπροσωπούσαμε τις τέσσερις βασικότερες πολιτικές ε, ομάδες ε, που είναι δραστήριες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποστηρίζουν ιδιαίτερως κάτι τέτοιο. Ενώ το δεύτερο θέμα ήταν η πιθανή εξέλιξη γεγονότων ε, και η επικύρωση το ε, συμφώνου εισδοχής το οποίο έχει ε, συμφωνηθεί μεταξύ ε, της Ουκρανίας αλλά και της υπόλοιπες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ ε, σημαντική ήταν η συνεισφορά του κυρίου Βαν Μπάλεν από την αποστολή μας, ο οποίος βοήθησε στην όλη ε, διαδικασία ε, για την Ολλανδική κυβέρνηση αλλά και τις Ουκρανικές αρχές. Το τέλος, όπως πάντα, ήταν ε, κλασικά ε, το να αποτίσουμε φόρο ε, στα θύματα της επανάστασης του Μαϊντάν. Ανάψαμε κεριά. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Οι περισσότεροι εξημών είμαστε τακτικοί επισκέπτες στο Κίεβο και την Ουκρανία αυτή λοιπόν ήταν η ενημέρωση. Δυστυχώς ε, άλλα μέρη δεν μπορούσαν να ε, συμμετάσχουν λόγω των ε, πτήσεων που είναι δύσκολες σήμερα. Ε, υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτές που θα ήθελαν να παρέμβουν. Κύριο Σετίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερος το ότι πήγατε μέχρι το Κραματόρες και, και ανατολικά του Δνύπερου. Ο Αντρί Πλένκοβιτς πριν από λίγες εβδομάδες έκανε ως μία από τις τελευταίες καλές πράξεις του πρωτού αποχωρήσει συμμετείχε στην οργάνωση της επίσκεψης αντιπροσωπείας στην Ουκρανία που υποτίθεται ότι θα πήγαινε στην, ε, ε, στα δυτικά του Ντονιέσκ, στη Μαριόπολη. Και τρεις-τέσσερις μέρες πρωτού γίνει το ταξίδι, μάθαμε από τον πρόεδρο Σούλτς και το επιτελείο του ότι δεν έπρεπε να διεξαχθεί η αποστολή διότι κινδύνευε η ζωή των βουλευτών. Τρεις αφάσαν παρόλα αυτά να πάνε, γιατί είχαμε κάνει όλη αυτή τη συνεργασία με τα μέλη του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Ως προεργασία. Και φυσικά δεν δέχτηκαν αυτή την ε, δικαιολογία και είπαν ε, ε, διότι χιλιάδες παιδιά ζουν σε αυτή την περιοχή και απερίψαν αυτή την αιτιολόγηση. Μάλλον το Προεδρείο του Κοινοβουλίου δεν θέλησε να ενοχλεί στο Κρεμλίνο. Και δυστυχώς ε, ε, ε, γίνεται συχνά αυτό, υποβαθμίζεται η κατάσταση. Βρίσκουμε δικαιολογίες για να μην ενοχληθεί η Ρωσία. Έχω πάει πάρα πολλές φορές στην Ουκρανία, στον Ντομπάς, 7 φορές. και κοντά στη Μαριούπολη ε, πολεμούν ακόμη ε, με πολύ μεγάλη γενναιότητα οι άνθρωποι και μην ξεχνάμε ότι υποστηρίζουν, υπερασπίζονται συγγνώμη και την Ευρώπη, όχι τη χώρα τους. την κυρία Αντρικίνα. Ευχαριστώ. Και πρώτα σας ευχαριστούμε για το debriefing για την κατάσταση. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τους πρόσφυγες. 1,5 εκατομμύριο ε, πρόσφυγες από την Ανατολική Ουκρανία έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φυσικά έχουμε και ηλικιωμένους και παιδιά μεταξύ αυτών. Πολλά δημοσιεύματα μιλάνε για την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το θέμα το γύρατε στις επαφές σας με τους υπουργούς ή μήπω μπορέσετε να πάτε σε κέντρα καταγραφής προσφυγών. Θα με ενδιαφέρει να μάθω αν έχετε στοιχεία. Γιουρέκ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που έγινε αυτή η αποστολή. Οι εταίροι μα από το Κοινοβούλιο και από τα κόμματα της Ουκρανίας τι πιστεύουν για την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ και ποιες είναι οι προσδοκίες τους από εμά. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. έκανα την ενημέρωση κυρίως για την αποστολή. Και για την αποστολή θα έλεγα ότι αυτό που έλειπε ήταν το περιεχόμενο των συζητήσεων. Δεν αναφέρθηκα σε αυτές. Εκτός από το θέμα της απελευθέρωσης, υποχρέωση θεωρήσεων και της επικύρωσης συμφωνίας σύνδεσης, διότι σίγουρα Πρωτίστως το έθεσαν οι Ουκρανικές αρχές αυτό το θέμα. Και τόνισαν ότι στην τρίτη επέτειο του Μαϊντάν είναι πολύ σημαντικό να είναι θετικό το μήνυμα που περνάμε στην κοινωνία των πολιτών. Και όλοι συμφωνήσαμε. Θυμούνται οι βουλευτέ από Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σίγουρα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο σημαντικό ήταν σε όλα τα στάδια αυτή τη διαδικασία να επιδεικνύουμε θετικά αποτελέσματα ε, γιατί αλλιώς ε, υπάρχει ε, μία κούραση και απογοήτευση, ε, λήψη πρόοδου. Σκληρές ε, μεταρρυθμίσεις έχουν επιβληθεί στην κοινωνία και έγιναν δεκτές από τους πολίτες με πρόταγμα την ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας της χώρας από σχέση με την εξωτερική απειλή υπό το μανδύα ε, των αποσχιστικών ε, κινημάτων. Ε, οι διοικητές των στρατιωτικών μονάδων μας έδωσαν στοιχεία και πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για τακτικούς στρατιώτες και και μέλη των αποσχιστικών αυτών ε, κινημάτων. Όντως, ήταν πολύ καλό που πήγαμε στην Ανατολική Ουκρανία και δεν είμαι η μόνη που το ζήτησα και πίεσα. Η γραμματεία το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό και ευχαριστώ τη γραμματεία. Μπορέσαμε να κάνουμε και επικοδομητικές συζητήσεις ε, και με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Το πλευρά του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας θεωρήθηκε φυσικά πάρα πολύ αρνητικό που δεν μπόρεσε η αντιπροσωπεία να μεταβεί στα ανατολικά της Ουκρανίας μετά από όλες αυτές τις ε, προετοιμασίες ε, των εθνικών βουλευτών. Και γι' αυτό και ικανοποιήθηκαν από την έκφραση της δικής μας αποστολής. Πάρα πολύ σημαντικό που είχαμε αυτές τις επαφές και για να απαντήσω στην κυρία Ανδρικίνα. Εσωτερικά εκτοπιστέντες ε, συναντήσαμε, αλλά όχι στα κέντρα ε, καταγραφής τους. Και είναι και πυκνό το πρόγραμμα για τα πολιτικά θέματα, αλλά και τα θέματα ασφαλείας δεν είναι εύκολο να πάει κάποιος ε, στα ανατολικά της Ουκρανίας. Μέχρι να φτάσουμε με αυτοκίνητο στο κραματός χρειάστηκε χρόνος. Ε, στον Ήπερο έπρεπε να πάμε με το αεροπλάνο. Ε, και ε, σκεφτήκαμε καταστάσεις ε, ε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ε. και στο κράματος ένα από τα σημεία της μερίσιας διάταξης ένα θέμα ήταν επαφές ε, με όλους εκπροσώπους ε, των ε, ΜΚΑΠΑΟ μικρών που βοηθούν τους εσωτερικά εκτοπιστέντες. Το συζητήσαμε. η κοινωνία των πολιτών αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα όπως αυτό της κοινωνικής ασφάλισης Υπήρχε μια σάφια σε σχέση με το καθεστώς ως προς την κοινωνική ασφάλιση δηλαδή των ε, εσωτερικά εκτοπιστέντων. Και υπάρχει το θέμα της επόμενης δεώσης του δανείου της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Ουκρανία που χρηματοδοτεί αυτό το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από ό,τι κατάλαβα. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, νομίζω ότι είναι ε, περίπλοκο το ζήτημα διότι δεν μόνο οι δημοσιονομικοί περιορισμοί το πρόβλημα. Ακόμη και χωρίς ε, τις συγκρούσεις, ακόμη χωρίς την επίθεση, ακόμη ε, και χωρίς την ανάγκη ε, άμυνας ε, ε κατά αυτής εξωτερικής απειλής υποκανονικές συνθήκες διακυβέρνησης, ε, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να εγκατασταθούν σήματα κοινωνικής ασφάλισης και όταν μιλάμε για εσωτερικά εκτοπιστέντες, πώς να γίνει έλεγχος. Υπάρχει αυτό το κενό η έλλειψη παραστατικών και τεκμηρίων για την πρόσβαση στο, στις κοινωνικές παροχές. Η κυβέρνηση αναγνώρισε το πρόβλημα και εδώ μπορώ να σας μιλήσω εξ για την, ε, τον έλεγχο ε, των ε, παροχών κοινωνικής ασφάλισης. περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι από το κράτος. Έχουν κάποια κατοχυρωμένα δικαιώματα. Όμως, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα πως ε, περιορίζεται σε ανθρωπιστική βοήθεια ή οποιαδήποτε, ε, οποιασδήποτε άλλη μορφής βοήθεια ε, παρέχεται τελικά στους εσωτερικά εκτοπιστέντες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να έχουμε επίγνωση όμως του ύψους των προκλήσεων στις οποίες ε, καλείται αυτή η κυβέρνηση να αντεπεξέλθει. Αυτή την εξήγηση θα σας έδινα. Ξέχασα κάτι μήπως. Σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις μου. Ο κύριος Πρέσβης ίσως θέλει να μας μιλήσει για την Ουκρανία. Please. Just press. Αναμφίβολα, η Ουκρανία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη διπλή κρίση, γιατί αφενός η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο στα εδάφη της Ουκρανίας και η στρατιωτική υποστήριξη που έλαβε η Ουκρανία από τη Δύση, παρόλο το μνημονίο της Βουδαπέστης, ήταν μεν πραγματική, αλλά πολύ περιορισμένη. Και οι Ουκρανοί απέδειξαν πως έχουν ένα πάθος για τη μάχη αυτή, οπότε μέσα στους περιορισμούς που έχουμε σε αυτό το πόλεμο με τη Ρωσία, έχουν δώσει τη μάχη και έχουν καταφέρει να φέρουν την κατάσταση σε μια ισορροπία δεν κατάφεραν να προχωρήσουν οι Ρώσοι, αλλά είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση 25 χρόνια διαφθοράς και κακής διακυβέρνησης. Και η κυβέρνηση σήμερα είναι μια μεταβατική κυβέρνηση όπου οι ηγέτες της ήταν πολύ άνετοι με την προηγούμενο καθεστώς, ξέρουν πως χρειάζεται να μεταρρυθμιστούν, να αλλάξουν, να αντιμετωπίσουν την διαφθορά και πιέζονται να το κάνουν από μια πολύ ε, ζωντανή και πολλά υποσχόμενη κοινωνία των πολιτών. Κάποιοι από την κοινωνία των πολιτών είναι υπουργοί, άλλοι υφυπουργοί, άλλοι μέλη του Κοινοβουλίου και πιέζουν την ηγεσία τους να κάνει τις σωστές επιλογές. Θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση και να πούμε πως Παρόλο που επιμένουν, επιμένουμε πως πρέπει να κάνουν σοβαρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως ε, μέχρι σήμερα η απόδοσή τους δεν ήταν κακή. Δεν ήταν εξαιρετική, αλλά έχουμε δει πιο ε, σοβαρές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια στην Ουκρανία από ό,τι είχαμε δει τα περασμένα 23 χρόνια. Και υπάρχει λόγος σοβαρός λόγος να είμαστε αισιόδοξοι πως θα τα πάνε καλά με τις μεταρρυθμίσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ εξοχότητα. Ήταν πολύ σαφές και εγώ συμφωνώ μαζί σας και πρέπει να πω πως πως ευχαριστώ τις Ουκρανικές αρχές γιατί μας πρόσφεραν την ασφάλεια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αποστολή και εμείς και η Συμβουλή μας και η Γραμματεία. Και πρέπει να σου πω πως ήταν απίστευτο, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Κραματόρσκ είχαμε τις μονάδες Α, οι οποίες μας συνόδευσαν και αισθανόμουν απολύτως ασφαλής. Ήταν πραγματικά εξαιρετική στη δουλειά τους. Um, Νομίζω πως ε, Μία ερώτηση ξέχασα να απαντήσω για τη συμφωνία του Μίνσκ. Ξέρουμε πως δεν είναι ιδανική η συμφωνία αυτή. Σίγουρα όμως οι Ουκρανικές αρχές είναι αφοσιωμένες στο να εκπληρώσουν την ε, συμφωνία αυτή και σε γενικέ γραμμές καταγγέλουν τις σοβαρές παραβιάσεις. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε και με άλλους ε, ε, εταίρους μας, για παράδειγμα με τους αξιωματούχους του ΑΣΕ που αναφέρονται στο θέμα αυτών των παραβιάσεων. ένα πολύ σημαντικό θέμα και το στο οποίο θα έπρεπε ενδεχομένω να σταθούμε παραπάνω σε μια επόμενη φορά είναι πως οι τεχνικές ικανότητες στα ανατολικά τμήματα της Ουκρανίας έτσι ώστε να καταφέρνουν να στέλνουν προπαγάνδα στις στις δυτικές, στα δυτικά τμήματα της Ουκρανίας, η εκπομπή δηλαδή σε τεχνικό επίπεδο που εκπέμπουν ενημέρωση και προπαγάνδα, τι να σας πω, δεν είναι συγκρίσιμο, γιατί οι δυνατότητες που είχαν για εκπομπή ε, των αυτονομιστών ήταν ε, απίστευτες και μου το είπαν αυτό και από τις μονάδες αιτιό, το οποίο για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Καλό είναι να το σκεφτούμε και αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και με το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Να σας ευχαριστήσω και τον πρέσβη κύριο Τζον Χάρστ. και για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Να σας πω ότι σας ευχαριστώ για όσες προφορίες μας δώσατε, για ε, την Κεντρική Ασία και την Ανατολική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Μεγάλη τιμή για μένα που βρέθηκα εδώ. Τώρα για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και για την κατάσταση της ασφάλειας εκεί θα διαπιστώσετε πως η Ευρώπη και η ΕΠΑ αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα είναι το πρόβλημα ε, του αναθεωριστικού Κρεμλίνου, ρεβιζιονιστές του Κρεμλίνου πια σήμερα. Και αυτό αποτελεί την πιο σημαντική απειλή και τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση σε επίπεδο ασφάλειας σήμερα. Γιατί τα λέω αυτά. Τελευταία 25 χρόνια μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει και να πούμε ότι είχαμε την πιο σταθερή και ευήμερη και σταθερή περίοδο ευημερία σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Παρόλε τις κρίσεις και τις τίτλους και τις επικεφαλίδες δεν είχαμε μεγάλους πολέμους και όταν μιλάω για μεγάλους πολέμους μεταξύ υπερδυνάμεων και θα σας το πούνε οι κοινωνικές επιστήμες ήταν η πιο ειρηνική περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εμείς επίσης διαπιστώσαμε που σημειώθηκε τεράστια αύξηση της ευημερία. Στα τέλη το 1990, στα τέλη του ψυχρού πολέμου, το 35% του πληθυσμού της γης ζούσε σε ε, μεγάλη φτώχεια. Το 2013 είχε πέσει στο 11% το ποσοστό αυτό. Ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας και γι' αυτό μιλάω για το θέμα αυτό, είναι η σταθερότητα στην Ευρώπη. Οι δύο πιο καταστροφικοί πόλεμοι στην ανθρώπινη ιστορία ήταν οι παγκόσμιοι πόλεμοι 1 και δύο που ξεκίνησαν και οι δύο στην Ευρώπη. Η παγκόσμια οικονομική τάξη, η οποία δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το δυτικό κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή η Παγκόσμια Τράπεζα, ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ΓΚΑΤ και μετά ο ΠΟΕ, ίδρυσαν ένα σύστημα οικονομικής ανάπτυξης που επέτρεψε σε κάθε χώρα στον κόσμο να ευημερήσει. key moment was the end of the Cold War. Και το σημείο κλειδί ήταν βέβαια το τέλος του ψυχρού πολέμου. Γιατί ήταν μεν ψυχρός ο πόλεμος αυτός και όχι καυτός, αλλά και πάλι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνος και είχαμε πάντα την απειλή μιας επικείμενης πυρηνικής, ενός επικείμενου πυρηνικού επεισοδίου και τι στήσαμε μετά τον ψυχρό πόλεμο ένα σύστημα ένομης τάξης και σύστημα ασφάλειας ε, μετα τον ψυχρο ενα συστημα ενομης ταξης και συστημα ασφαλειας μετα ψυχροπολεμικο που βασιζόταν στις εξής αρχές. Κυρίαρχα εθνικά κράτη σε ασφαλή σύνορα με τη δυνατότητα να επιλέξουν τα ίδια την τύχη τους βασιζόταν στην αρχή πως ο πόλεμος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως τρόπος για να επιλύονται ζητήματα μεταξύ κρατών. Η ειρηνική επίλυση διαφορών. Και στην ψυχροπολεμική περίοδο έγινε μια μεγάλη οικοδόμηση θεσμών στην Ευρώπη, επέκταση και διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και αυτή η διεύρυνση δεν έγινε υποχρεωτικά, δεν ζητήσαμε από τους γείτονες να ενωθούν μαζί μας. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκαναν προσπάθειες για να έρθουν οι όμορες χώρες να συνταχθούν μαζί τους. Ήταν η ελεύθερη βούληση των νέων κρατών αυτών και των θεσμών που αισθάνθηκαν να τις προσελκύουν τα ιδανικά και η ευημερία αυτών των οργανισμών. Αυτών των δυτικών οργανισμών είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι χώρες αυτές έπρεπε να γίνουν δημοκρατίες, να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η διαφθορά, να φέρονται στις μειονότητες τους με ανθρώπινο και δίκαιο τρόπο. Για παράδειγμα, τα προβλήματα των μειονοτήτων που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χρειάστηκε να επιληφθούν και έγινε αυτό. δυστυχώς αποδείχθηκε πως δεν δέχτηκαν όλες οι χώρες αυτή την μεταψυχροπολεμική τάξη. Και μπορεί να πει κανείς ότι αν δούμε πέραν των τελευταίων οκτώ ετών αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως η κυβέρνηση της Ρωσίας δεν δέχεται αυτή την κατάσταση. Έχουμε αξιωματούχους της Ρωσίας που το ξεκαθάρισαν τόσο πολλές στιγμές λέγοντας πως η Ρωσία θα πρέπει να έχει σφαίρα επιρροής. Και αυτή η σφαίρα επιρροής αυτή τη στιγμή είναι κατελάχιστον τα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και με κάποιες ερμηνείες συμπεριλαμβάνει και το πρώην σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και είπαν απερίφραστα και όποιος πήγε στο Βαλτάι είπαν πως η παγκόσμια τάξη νέοι κανόνες ή καθόλου κανόνες. Οι κανόνες που θέλουν να αλλάξουν είναι οι κανόνες της περίοδου της μεταψυχροπολεμικής. Ο κύριος Πούτιν πολλές φορές δήλωσε και το έκανε και ο κύριος Λαυρόφ και άλλοι εξωματούχοι πως η Ρωσία έχει το δικαίωμα και μάλλον το καθήκον να προστατεύει τους ε, κατευθυνότητα Ρώσους και τους Ρωσόφωνους όπου και, όπου και αν ζουν. Also, look carefully. Επίσης, αν εξετάσει τις δηλώσεις περί εθνικής κυριαρχίας θεωρούν πως μόνο τα πολύ ισχυρά κράτη είναι ε, πραγματικά κυρίαρχα και όλοι οι υπόλοιποι έχουν ένα μικρότερο βαθμό εθνικής κυριαρχίας από ότι τα ισχυρότερα κράτη. Αν αυτό είχε να κάνει μόνο με ρητορική που απευθύνει το Κρεμλίνο, δεν θα μας ανησυχούσε ιδιαίτερα. Αλλά αν δείτε την τάση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής για τα τελευταία 9-10 χρόνια, ναι, υπάρχει λόγος ανησυχίας. Να ξεκινήσουμε κατελάχιστον μετά, την, ε, μετά τον κυβερνοπόλεμο κατά της Εστονίας το 2007, κυβερνοπόλεμος που ξεκίνησε και καλυμμένα βέβαια από τη Ρωσία. Και γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί οι Εστονοί κατέβασαν ένα μνημείο που είχε στηθεί για να εορτάσει την ε, ενσωμάτωση μέσω κόκκινου στρατού της Εστονίας στη Σοβιετική Ένωση. Μετά είχαμε τον πόλεμο κατά της Γεωργίας, που θεωρητικά έκλεισε το καλοκαίρι του 8. Αλλά αν διαβάσετε πριν από ένα μήνα του New York Times θα δείτε πως η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της Νοτιού Ασετίας και της Απχαζίας αφενός και της υπόλοιπης Γεωργίας από την άλλη μετακινείται μερικά μέτρα κάθε δύο μήνες και τρώει και άλλα κομματάκια της γεωργίας. Και μετά βέβαια είχαμε και την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία, μια προσάρτηση από ρωσικά στρατεύματα και μετά και τον Ιβριδικό πόλεμο που ξεκίνησε στην περιοχή του Νταμπά στο Κρεμλίνο σύντομα μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Has been slow to react to this even after the annexation of Crimea. Και μετά την προσάρτηση, να σας πω πως άρχισαν τα προβλήματα της Ανατολικής Ουκρανίας. Ξέρετε πως πολλοί κόσμος έπαψε να θέλει να περιγράφει αυτό που συνέβη στην Κρυμαία ως ε, στρατιωτικό πραξικόπημο από το Κρεμλίνο. Και το είδαμε στην περιγραφή που έγινε και στην Ανατολική Ουκρανία, που το λέμε εμφύλιο πόλεμο, που είναι αδιανόητο. Αυτό ήταν ένα πόλεμο, τον οποίο σχεδίασε χρηματοδότησε, του οποίου ηγήθηκε, εξόπλησε και ε, υποβοήθησε η ρωσική πλευρά στέλνοντας δε και ρωσικά στρατεύματα. Τι έγινε, ε, είχαμε την κατάρριψη του αεροπλάνου της Malaysia Airlines όπου η Δύση δεν θέλησε να δεχτεί πως ήταν πύραυλος Μπούχ από τους Ρώσους που έκανε την κατάρριψη. Και ήτανε Ρωσοί στρατιώτες ή οι στρατιώτες με στήριξη της Ρωσίας που έστειλαν αυτό τον πύραυλο. Οπότε δεν θέλουμε να δεχτούμε ε, αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι στοιχεία πιστικά, πως θέλει να αναθεωρήσει την τάξη, τη μεταψυχρομολυμική τάξη πραγμάτων, το Κρεμλίνο. Και θέλω να σας πω πως αυτό δεν θα τελειώσει στην Ουκρανία. Και κάποιες φωνές στην Ευρώπη και κάποιες φωνές στη ΣΥΠΑ δέχονται αυτή την προπαγάνδα του Κρεμλίνου. Και λένε πως η Κρυμαία ήταν μια μοναδική περίπτωση. Και αν απλώς αποστρέψουμε το βλέμμα και αφήσουμε τη Μόσχα να αποστηθεροποιήσει την Ουκρανία, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για περαιτέρω επιθετικότητα του Κρεμλίνου. Αυτό είναι ευχολόγια και είναι οι ανώτατοι αξιωματούχοι που λένε πως οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν ε, το Κρεμλίνο να παρέμβει στην Ουκρανία και να ξεκινήσει αυτό το πόλεμο ισχύουν και για άλλες περιοχές. Η ρωσική αρχή, και το λέω αυτό συσσαγωγικά, της υπεράσπισης των εθνικών μειονοτήτων και των ρωσόφωνων έχει να κάνει με τη Λετωνία. 25% του πληθυσμού μπορεί να περιγραφεί με αυτόν τον τρόπο. Στην Εστονία 25% έτσι μπορούν να περιγραφούν στο Καζαχστάν. Μιλάμε για την Κεντρική Ασία. Εκεί έχουμε πάλι 25% του πληθυσμού που περιγράφεται ως ρώσικη μειονότητα ή ρωσόφωνη και στο Καζαχστάν. Ο πληθυσμός αυτός βρίσκεται στα βόρεια σύνορα με την Ρωσία, στην περιοχή που έχει πάνω από από τρίτα των υδρογονάνθρακων ε, της χώρας. Το καλοκαίρι του 2004 στην λίμνη Ζέλικο όπου συναντιόνται τον Αύγουστο ε, όλοι οι Ρώσοι ηγέτες με τη ρωσική νεολαία ο κύριος Πούτιν μίλησε για το Καζαχστάν ως τεχνητή χώρα. Είπε πως ο φίλος του πρόεδρος Ναζαρμπάγεφ ήταν πραγματικά πολύ εφευρετικός. Είναι ε, μεγάλο πνεύμα που κατάφερε να δημιουργήσει αυτό το τεχνητό κατασκεύασμα. Και φέρεται πολύ σωστά στους Ρωσόφωνους και στους Ρώσους. Αλλά όπως είπε ο κύριος Πούτιν δεν ξέρουμε πώς και τι θα ακολουθήσει. Προτείνω πως όποιος νομίζει πως ο κύριος Πούτιν κλείνει τις φιλοδοξίες του στην Ανατολική Ουκρανία θα πρέπει να συγκρίνει τόσο είπε στη Λίμνη Ζέλικο για το Καζακστάν με τα όσα είπε στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο, Σύνοδο του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία. Στον πρόεδρο Μπούστα είχε πει. Ήθελα να πω τα εξή. Ο κύριος Πούτιν έχει φιλοδοξίες που ξεπερνάνε την Ανατολική Ουκρανία και πέραν της ε, σφαίρας επιρροής στην Ανατολική Ουκρανία. Θα ήθελε να υποσκάψει το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει νέους κανόνες παιχνιδιού στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία που δεν συμφωνούν με τις αρχές μας, με τις αξίες μας και με τα συμφέροντά μας. Και το βλέπω αυτό όχι μόνο στα λιγόμενά του για το, για το Καζακστάν, αλλά το διαπιστώσαμε την ημέρα που έκλεισε το 2014 η Σύνοδος ΝΑΤΟ ε, στην Ουαλία. Και δύο μέρες μετά που πήγε ο πρόεδρος Ομπάμα στο Τάλιν για να τους ε, επιβεβαιώσει πως αν γίνει επιθετικό το Κρεμλίνο η Δύση θα τους στηρίξει τους Εστονούς. Και την ημέρα που τελείωσε η σύνοδος αυτός, το Κρεμλίνο απήγαγε από την Εστονία έναν ε, μυστικό πράκτορα έτσι ώστε να μην ε, έχουν καμία δυνατότητα παρανόησης οι κάτοικοι της Βαλτικής στο τι συμβαίνει. Ε, απήγαγαν και έναν ε, Λιθουανό από την ε, Βαλτική θάλασσα 15 μέρες αργότερα. Είναι πολύ γνωστή η στόχη, όχι μόνο να επεκταθεί η Ρωσία, αλλά και να υποσκάψει τους θεσμούς που δημιουργήσαμε στην Ευρώπη, τους οποίους δημιουργήσαμε για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα. Και γι' αυτό οι χώρες, οι βόρειε χώρες αυτή τη στιγμή κάνουν μια συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και είναι οι προκλήσει του Κρεμλίνου οι οποίες έχουν ξεπεράσει ακόμα και την ευρύτερη ε, σφαίρα επιρροή που ήταν, αν όχι οι πρωινέ, είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, γιατί φτάσανε τα υποβρύχια ε, στα ύδατα της Σκανδιναβίας, είδαμε βομβαρδιστικά που έφτασαν πολύ κοντά σε ε, αεροπλάνα του ΝΑΤΟ ε, που ε, κλείνουν τους πομπούς έτσι ώστε να μην γίνει έτσι ώστε ενδεχομένως να σημειωθεί επεισόδιο και μην σας κορυδεύουν από τη γραμμή του Κρεμλίνου ότι όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Μη σας κορυδεύουν. Τι κάνει αυτό που κάνει η Μόσχα στην Ουκρανία, που συνεχίζει να κάνει στη Γεωργία, είναι να χρησιμοποιεί μια τακτική των παγωμένων σειράξεων. Οι παγωμένες σειράξεις τι σημαίνουν. Όπου υπάρχουν εθνικές διαφορές και όπου υπάρχουν ε, ε ρωσόφωνοι και ρώσικες μειονότητες θα χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσει περισσότερη επιρροή στις χώρες στις οποίες βρέσκονται η Ρωσία. Η Σοβιετική Ένωση καταλήθηκε το 1991 και την επόμενη μέρα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Αμήνης και δεν ξέρω αν αυτό είχε την έγκριση του τότε πρόεδρου Γέλτσεν, ακολούθησαν αυτή την τακτική του μοντέλου των παγωμένων σειράξεων στον Αγκόρνη Καραμπάχ, στο Αζερβαϊτζάν δηλαδή, στην Απχαζία, στην Νότια Οσετία, στη Γεωργία, στο, στην Υπερδνηστερία, στη Μολδοβία. Και αυτό είχαμε δύο χρόνια πριν οποιοδήποτε μιλήσει για διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Η τακτική αυτή είχε ήδη χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται και σήμερα στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει πολύ πριν διευρυνθεί το ΝΑΤΟ και πολύ πριν διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και να μην, και να μην παρασυρώμαστε από σιρήνες που λένε πως η Δύση δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Αν αφήσετε ελεύθερο χώρο ε, ελιγμών στον Πούτιν στην Ουκρανία, σας εξασφαλίζω πως θα έχετε προβλήματα αλλού. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις ε, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Ε, προσφάτως είχαμε ε, τις προεδρικές εκλογές και σίγουρα πρέπει να αναφερθώ στην επιρροή των εκλογών αυτών για τα αποτελέσματα και την επιρροή που θα έχουν στην ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Έχουμε έναν ντολοδόχο πρόεδρο ο οποίος έχει πει ε, διάφορα πράγματα για ε, το ΝΑΤΟ, για την ε, Ρωσία και την Ουκρανία. Ισχύει επίσης ότι είπε διάφορες, υπέπεσε σε διάφορες αντιφάσεις για αυτό και πολλά από τα σχολεία του δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι πολίτες ανησυχούν για την δέσμευση των ΙΠΑ στο ΝΑΤΟ και την στάση ε, που θα έχει απέναντι σε αυτό ε, το ε, ρεβιζιονιστικό Κρεμλίνο. Ανησυχώ, καταλαβαίνω αυτές τις ανησυχίες και δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του εντελοδόχου Προέδρου Τραμπ, όμως νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος από ό,τι νομίζουν πολλοί. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό δεν ξέρουμε αν αυτά τα οποία είπε ο ε, Τραμπ ε, είναι αυτά τα οποία θα τηρήσει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Ισχύει όμως ότι υπάρχουν ομάδες ε, στην ομάδα του που έχουν ξεκάθαρες απόψεις όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ΝΑΤΟ, την, την ανάγκη να σταματήσουμε τη Ρωσία, την αναθεωριστική ε, την Ρωσία ε, και την περίπτωση πολέμου ε, κατά της ε, δεύτερης μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης του πλανήτη. Ο αντιπρόεδρος Πένς έχει μια σταθερή στάση για αυτό και όσοι έχουν ακούσει την, τον debate των αντιπροέδρων γνωρίζει τι έχει να πει για όλα αυτά. Δεν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Φλίν αλλά ε, και οι ε, θέσεις ε, της Katie Μερφάρλαντ είναι ξεκάθαρες. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών, όμω τα ονόματα τα οποία αναφέρθηκαν είναι ο Ρούντι Τζουλιάνι, Μιτ Ρόμνι, ο κύριος Πετρέας. Όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί πάνω σε αυτό το ζήτημα. και το όνομα το οποίο συζητάτε προσφάτως ε, Μάντισον ε, για, την, ε, για το Υπουργείο Αμήνης είναι επίσης πολύ καλό. Εάν ο κύριος Τραμπ κατευθυνθεί προς την λάθος κατεύθυνση για να έχει μια πιο φιλική σχέση με τον Τραμπ, τότε υπάρχει, με τον ε, Πούτιν, τότε υπάρχει ένα ε, προστατευτικό τείχος ε, στη Σύγκλιτο. Υπόθηκε ότι θα ήταν λάθος ε, να αλλάξουμε την πολιτική μας απέναντι στην Ρωσία και την Ουκρανία. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να υψώσουμε το ανάστημά μας σε έναν μπούλι στο Κρεμλίνο. θα αποτελέσει έκπληξη για μένα στην περίπτωση που ο Τραμπ κατευθυνθεί προς τη λάθος κατεύθυνση διότι θα έχει μια δύσκολη μάχη από το Κογκρέσο και σε περίπτωση που τον Μάρτιο όταν θα πρέπει να ανανεώσει τις κυρώσεις αν αφήσει να χαλαρώσουν Σε περίπτωση λοιπόν που χαλαρώσει τις κυρώσεις, τότε υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσει νομοθεσία από το Κογκρέσο που θα επιμείνει ε, για αυτές και νομίζω ότι θα υπάρχει υποστήριξη και από ε, τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ασκηθεί και βέτο. Όποιος γνωρίζει την Αμερικανή εξωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ε, γνωρίζει τι συνέβη τη δεκαετία του 70 ε, ο οποίος ε, είχαμε έναν Υπουργό Εξωτερικών ε, Jackson Φάντικ ο οποίος δεν ήθελε να δυσχεραίνει την κατάσταση και τότε ακολούθησε βέτο από τον Κογκρέσο. Σίγουρα θα, είναι ένα πολιτικό, θα υπάρξει πολιτική επέμβαση για τον κύριο Τραμπ σε περίπτωση που κατευθυνθεί προς τη λάθος κατεύθυνση. Και μερικά τελευταία σχόλια θα ήθελα να σας πω τις ε, προτάσεις, ε, τις πολιτικές προτάσεις που σίγουρα περιμένετε, αλλά θα τις παρουσιάσω παρόλα αυτά. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό κίνδυνο, ο οποίος απαιτεί μια σοβαρή απάντηση. Οι στόχοι του κυρίου Πουτίν ξεπερνούν την περιοχή της ε, Έσουσουδού το που περιλαμβάνει ε, τρεις συμμάχους του ΝΑΤΟ και πολύ πιθανό να ξεπεράσει αυτά τα όρια και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια αυστηρή πολιτική για να τον αποτρέψουμε να λάβει περαιτέρω βήματα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε θέματα. Η σύνοδος ε, της ε, Βαρσοβίας ήταν ξεκάθαρη, ούτως ώστε να θέσει στρατιωτικές ομάδες ε, στην, ε, στις χώρες της Βαλτικής και η απόφαση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια αυστηρότερη πολιτική ε, ε, από την πλευρά του ΝΑΤΟ και τη στάση των ρωσικών ε, αεροπλάνων προς τα πλοία του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα επίσης να δω πιο αυστηρές κυρώσεις, το οποίο νομίζω θα είναι δύσκολο να προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως θα πρέπει να το συνεχίσουμε διότι ασκούν σοβαρέ οικονομικές ποιώσεις, διότι σύμφωνα με το ΔΝΤ αλλά και ανώτατα στελέχη οδηγούν σε μείωση 1,5% του και γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν θέλει απεγνωσμένα να χαλαρώσουν αν όχι να καταργηθούν. Επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε περαιτέρω την Ουκρανία που θα πρέπει να είναι διτής μορφής. Πρώτον, περαιτέρω οικονομική υποστήριξη. Έχουν να αντιμετωπίσουν στην Ουκρανία δύο σοβαρές ε, προκλήσεις ε, ε, ε, έχουν έναν πόλεμο και από την άλλη έχουν την οικονομική ε, υποστήριξη των πολιτών. Ο Summers αναφέρθηκε για 10 δις τα οποία πηγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Ακούγεται ως κάτι αξιόλογο. Ο Λάρι το περιγράφει ως επένδυση στην ασφάλειά μας και έχει απόλυτο δίκιο με αυτό. Θα πρέπει να παράσχουμε επίσης περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Γνωρίζω ότι ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο είναι διφορούμενο. Δεν είμαι απεσιόδοξος όσον αφορά την πολιτική ε, του Τραμπ, όμως δεν ξέρω αν θα ήταν διαθέσιμος να το κάνει. Ελπίζω όμως ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα είναι διατεθειμένη να το κάνει και ελπίζω η Ευρώπη να το αποδεχτεί και να μην, το, ε, και να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Επίσης καταλαβαίνω ότι οι στόχοι του Πούτιν ξεπερνούν την Ουκρανία. Ίσως το Καζακστάν ακόμα θα πρέπει να τον σταματήσουμε και το μέρος για να σταματηθεί είναι η Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Θα ξεκινήσω με τα δικά μου σχόλια. Σύμφωνο. Με αυτά που είπατε, κυρίως στο τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής σας, εκπροσωπώ την Πολωνία. εδώ στο Κοινοβούλιο και είμαστε υπέρ της διαθλαντικής σχέσης, αυτό δεν είναι κανένα μυστικό. Και θέλουμε να συνεργαστούμε με όποια ε, αμερικανική κυβέρνηση είναι στην εξουσία. Παραμένουμε αισιόδοξη και θα ήθελα να σας πω ότι οι πολιτικές της Ρωσίας ήδη από το 2005 ήταν ξεκάθαρες ε, και αποτυπώνονταν σε έγγραφα πολιτικής και δόγματα ε, που εξέδωσε η Αμερικανική κυβέρνηση. Κατά πάσα πιθανότητα Το λάθος μας ήταν η έλλειψη ε, συνεκτικής ε, συμπεριφοράς. Ε, όταν μιλάμε για, ελέ, ε, για συστήματα αμοιβαίου ελέγχου, ε, αυτά τα περίφημα checks and balances, και αναφέρομαι στο 2009, και να επισημάνω ότι ο Κατζίνσκι, ο εκλειπών πρόεδρός μας ήταν, ε, μιλούσε και ευθαρσούσε αλλά ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό ε, στην αποτροπή τέτοιων ε, τάσεων από τη Ρωσία. Και σε το του 2007, στην αισθανική κρίση, αν θυμάμαι καλά, Τέλειο Απριλίου, αρχές Μαΐου, έτσι, 2007. Η Πολωνία ήταν αυτή που προσέφερε ε, πολύ ε, υποστήριξη προς την Εστονία που τη ζήτησε. Επίσης η Πολωνία και ο πρόεδρος καζίνσκι. το διαβούλευσης με ΣΥΠΑ και άλλοι ηγέτες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρενέβησαν τον Αύγουστο του 2007 στην Γεωργία, το 2008. Ποιο δίδαγμα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την κρίση. επαναξιολόγηση συμπερασμάτων ε, σε όλο και το δυτικό κόσμο, ε, η έκθεση του κυρίου Ταβίνη για τις ε, ε, ρίζες της κρίσης ήταν μια απλή αλληλουχία των γεγονότων από την κρίση ε, στην Αστονία και μετά στη Γεωργία. Πολλά γεγονότα παραμένουν αντιευκρίνιστα για πολλούς, ε, αλλά όχι για τους Πολωνούς και θα προσθέσω και το Σμόλενσκ σε αυτό. Αλλά σίγουρα σε αυτά συγκαταλέγεται και η προσάρτηση Κρυμαίας. Όταν υιοθετούμε μία ε, αποφασιστική στάση ενώπιον της Ρωσίας, όλο κάτι γίνεται σε επίπεδο διπλωματικής ε, δραστηριότητας. Υπάρχουν τα αρνητικά ζητήματα ε, ε σε σχέση με τη Ρωσία, την Ουκρανία και προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε με τα θετικά, ε, τις θετικές πτυχές της συνεργασίας μας. Και ξέρετε τι υπερτερήφ. Ναι, σας ξαφνιάζω το θετικό θεματολόγιο. Η Αρκτική, παραδείγματο χάρη. Θυμάμαι ακόμη την ε, συζήτηση στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη του 2015 μας μιλούσαν για την θετική έκβαση της παρέμβασης της Ρωσίας στη Συρία και νωρίτερα η πιθανή λύση των χημικών όπλων στη Συρία τι λείπει στο δημοκρατικό κόσμο, συνεκτικότητα και ξεκάθαρη σε παγκόσμιο επίπεδο διάγνωση των ε, προβλημάτων και των ζητημάτων. Ο κύριο Θετίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ναι, τα ακουστικά θα τα χρειαστείτε. Κυρίε και κύριοι. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ. Ήταν ε, περιστατωμένη και διεξοδική η, η εικόνα της Ρωσίας που παρουσιάσατε ως υπεραλιστικής δύναμης. να αναφερθώ σε αυτό ε, στο οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι. Συμφωνία Μίνσκ. Είπε, ε, υπόθηκε ότι ε, το τίμημα της συμφωνίας ε, με τη Ρωσία είναι αυτό του χαρτιού στο οποίο γράφεται η συμφωνία έχει, ε, ε, ήταν εθνισυγενής η συμφωνία και αν όχι έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Να ζητώ ένα εφεδρικό σχέδιο. Δεν λειτουργεί αυτή η συμφωνία. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα ρεαλιστικό με εναλλεκτικό σχέδιο χρειάζεται υποστήριξη, η Ουκρανία χρειάζεται στρατιωτικό υλικό, πυρομαχικά, όπλα για να μπορέσουν να μηνθούν οι Ουκρανοί. Ή μήπως, κύριε Πρέσβη, διαβλέπετε εσείς κάποια άλλη δυνατότητα για να πάψει η σύγκρουση. Να αποκατασταθούν τα εδάφη στην Ανατολική Ουκρανία. Κύριε Ανδρική, τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη. Πολύ ενδιαφέρουσα και ενθαρρυντική η παρουσίαση, θα έλεγα. Εγώ είμαι από τη Λουθανία. Νομίζω ότι αυτό σας προειδεάζει για αυτά που θα πω. Μιλήσατε για την περίοδο μετά το ψυχρό πόλεμο. Τα τελευταία 25 χρόνια ήταν τα πλέον ειρηνικά και σταθερά στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Σας θυμίζω όμως πως σε αυτήν την περίοδο ε, κατέρευσε το Σοβιετικό μπλοκ. Εγώ στις 9 Δεκεμβρίου, και μόνο εγώ και οι συμπολίτε μου, θα εορτάσουν 25 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας της ε, Λευκορωσίας από το Σουσκέβιτς, ε, από το Χρατσκούφ, ε, πλευρά της Ουκρανίας, από το Μπορις Γέλτσιν, πλευρά της Ρωσίας. Και δεν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση ειρηνικά διαλύθηκε εκ των όνων συνετέ, συνετέθη η υπερδύναμη. Στη Δύση έλεγαν οι ειδικοί ότι πρόκειται για καταρρεύση της Σοβιετικής Ένωσης και αυτό θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, θα προκύψουν νέες πυρηνικές δυνάμεις. Που δεν είναι καταστροφή για την Ουκρανία και ε, ε, κατόμβη για πολλές χώρες. Όταν υπεγράφει λοιπόν αυτή η συμφωνία, έλεγε πως η Σοβιετική Ένωση ως υποκείμενο ε, προσωπικότητα διεθνούς δικαίου δεν υφίσταται πλέον. Μπορώ να προσυπογράψω αυτά που είπατε για τις παγωμένες σειράξεις. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Χρειαζόμαστε εργαλεία δεν για να, αντιμα... Ε, για να αντιπαλέψουμε αυτή την ε, τακτική της Ρωσίας. Εγώ πιστεύω ότι οι κυρώσει, βασικότερο εργαλείο που έχουμε, πρέπει να είναι ισχυρότερε. Για να δείξουμε ότι δεν μας αρέσει αυτό που κάνουν στην Κρυμαία και στην Ουκρανία. Οι ε, πρόσωποι της δημοκρατικής ε, αντιπολίτευσης ε, στη Ρωσία πιστεύουν ότι είναι πραγματικά αμεληταίο το αποτελέσμα των κυρώσεων που έχουμε επιβάλει. Για την Ουκρανία. Πρέπει να καταλήξουμε συμφωνίες στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διασυλλαντικό επίπεδο, διότι όταν ο νέος πρόεδρος στην προεκλογική του εκστρατεία μιλούσε για την Κρυμαία και έλεγε ότι πρέπει να, είναι, να ανήκει στη Ρωσία. Δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές αυτές οι δηλώσεις. Και μία ερώτηση. Την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο ε, το Ίδρυμα Μπόρις Νέμτσεφ ε, ε, ε, ε, διοργάνωσε ένα ε, βήμα για τις σχέσεις με τη Ρωσία και συζητήθηκε το θέμα για τις κυρώσεις. Κοντοκόψιο, ο, ο βασικός ομιλητής είπε πως αυτές οι κυρώσεις δεν είναι κατά του Κρεμλίνου αλλά τελικά πλήττουν τη Ρωσία για τους Ρώσους και είπε Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταλάβουμε τις μηχανογραφίες και την προπαγάνδα και πώς λειτουργούν οι κυρώσεις. Αλλά κάποια λύση σίγουρα πρέπει να βρεθεί. Ευχαριστούμε, friend. Ευχαριστώ. και παίζει. θέλω να προσεγγίσω το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία. Όταν σας άκουγα, ξεκάθαρα είχα την αίσθηση ότι ε, πώς να πω, έχετε κάποιο σκεπτικισμό σε σχέση με την, τον Τραμπ και την ικανότητα που έχει από την αρχή της θητείας ε, να αντιμετωπίσει την άλλη υπερδύναμη. Είπατε όμως ότι το NSA, το Υπουργείο Αμήνης, ε, ανώτατη σύμβουλη για θέματα άμυνας, θα τον ε, μαζέψουν ε, όταν πρόκειται να εφαρμόσει την πολιτική, ό,τι και αν έχει στο μυαλό του. Θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά θα έρθει η μέρα που θα πάει σε αυτή την αίθουσα που λαμβάνει τις στρατιωτικές αποφάσεις ο κύριος Τραμπ και Ξέροντας πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, πάντοτε υπάρχει διελκυστίδα ανάμεσα σε αυτούς ε, που θέλουν το ΜΕΝ και αυτούς που θέλουν το ΔΕ και διαφορές ανάμεσα στα Υπουργεία και στις διάφορες συναρμόδιες αρχές. Σε αυτό το Situation Room, λοιπόν, θα έχετε τη μία πλευρά που θα λέει άσπρο και την άλλη πλευρά που θα λέει μαύρο, θα λέει όχι δεν ε, νομίζουμε ότι είναι καλή ιδέα να γίνει αυτό και εσείς, Πρόεδρε, θα αποφασίσετε. Πώς αισθάνεστε άνετα εσείς όταν σκέφτεστε τέτοιες καταστάσεις που θα ανακύψουν α, ε, ε, ε, οπωσδήποτε, γιατί αναπόφευκτα, γιατί πάντοτε έτσι γίνεται. Δεύτερη ερώτηση και θα παραθέσω σύντομα ε, κάτι που υπόθηκε για την Ουκρανία. μετά από αυτή την, ε, τις δεκαετίες εκλεπτοκρατικής ελίτ ε, που ε, μετέτρεψε τη χώρα, φτωχοποίησε αυτή τη χώρα και μετά από τη ληστρική επιδρομή αυτών των διεφθαρμένων πολιτικών έχει μείνει χωρίς πλουτοπαραγωγικούς πόρους η χώρα. Ξέρετε ποιον παρέδεσα, τον Μιχαήλ Σακασφίλη που πριν από λίγες εβδομάδες ε, ήταν στην όδησό ε, ε, ε, κυβερνήτης και μίλησε για την διαφθορά λοιπόν, την ενδημική διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα να τροφοδοτήσουμε αυτή τη χώρα και με άλλα κονδύλια που ουσιαστικά θα ροκανιστούν από αυτούς τους ε, διεφθαρμένους αξιωματικούς ε, που ε, ληστεύουν συστηματικά τη χώρα. Ευχαριστούμε. Μάρικ Μήπως να ακούσουμε τις απαντήσεις του, του πρέσβη. Φοβούμαι ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για άλλες ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη για όσους ε, ήθελαν και να κάνουν και άλλες ερωτήσεις ε, και ευχαριστώ και τους που θα παραμείνουν ε. λίγο παραπάνω. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρέσβη. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε. για τι ευαλτικέ χώρε, για την Κεντρική Ασία και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μα είπε για το μέλλον. Εγώ θέλω να ρωτήσω για το παρελθόν. Πώ αποτιμάτε την ε, περασμένη δεκαετία Γιατί δεκαετία, διότι σωστά υπέδειξε η πρόεδρος μας πως εμείς που επισκεφθήκαμε τη Γεωργία Διαπιστώσαμε η δίσομαση ότι η σύραξη δεν ήταν παγωμένη. Ε, ακόμη και πριν το 2008 υπήρξαν επεισόδια. Ε, καταρρίφθηκαν ελικόπτερα και πριν από το 2008. Πώς αντίδρασε η Δύση. Τα τελευταία 10 χρόνια κρίνεται ικανοποιητικές αντιδράσεις της Δύσης. Τι είναι, επαναλαμβάνεται η κατάσταση του 39, η σύμμαχοι της ε, Πολωνίας εισήλθαν σε αυτή την ε, περίεργη περίοδο παρά την εισβολή ε, όπου δεν έκαναν τίποτα μέχρι να μπει ο Χίτλερ στην Ολλανδία. Μήπως να κάνουμε ένα παραλληλισμό. μήπως αυτή η απάθεια επηρεάζει την ε, ε, ισορροπία ε, του στρατηγικού σχετισμού δυνάμεων. Τι θα γίνει με τα ενεργειακά ζητήματα, το Nord Stream 2. Ξέρετε τι έγινε με το Nord Stream 1 για τις Βαλτικές χώρες και την Πολωνία. Και τώρα με το Nord Stream 2 θα, θα χάσει το καθεστώς χώρας διέλευσης για το φυσικό αέριο. Η Ουκρανία. Λοιπόν, από το 2008 κρίνεται ότι ήταν ικανοποιητική η αντίδραση για την ε, Ουκρανία και για τη Γεωργία. Δεν θα έπρεπε να έχουμε υποστηρίξει τη Γεωργία, δεν θα έπρεπε να έχουμε ε, προλιάρει τον δρόμο της Γεωργίας ε, προς το ΝΑΤΟ. Ακούσατε τι είπε ο Σακασβίλη. Δεν θα έπρεπε να έχουμε υποστηρίξει τις βαλτικές χώρες, τη Λετονία και την Εστονία. Ευτυχώς η Λιθουανία δεν απειλείται τόσο πολύ από γεωπολιτικής πλευράς. Όπως η Λετωνία και η Εστονία δεν κινδυνεύει τόσο πολύ. κρίνεται ότι είναι σταθερή κατάσταση. Ε, ε πώς αποτιμά την τελευταία δεκαετία, γιατί αυτό θα, προ, θα ε, προϊονίζει και το μέλλον. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει Πρόεδρος, αλλά έχουμε και χρονικούς περιορισμούς. Ζητώ συγγνώμη. Κύριος Πρέσβης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω γρήγορα κάθε μια ερώτηση που άκουσα. Συμφωνώ καταρχήν για το Plan B για την περίπτωση του Μίνσκ. Είναι μια συμφωνία που έχει πολλά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, γιατί δεν έχει προετοιμαστεί και συγγραφεί για να αποδείξει ότι υπάρχει θήτης και θύμα. Και είχαμε μία συμφωνία την οποία καταπάτησε το Κρεμλίνο που ήταν το Μίνσκ 1 και μετά τη Μίνσκ 2 η οποία ήταν πιο ευνοϊκή για το Κρεμλίνο και μετά υπεγράφει. Νομίζω όμως πως παρόλα αυτά, αν κάνουμε έναν απολογισμό, είναι θετικό γιατί είναι το όχημα μέσω του οποίου επέβαλε κυρώσεις και διατηρεί κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Οπότε παρόλε τι εγγενείς αδυναμίες του έχει χρησιμοποιηθεί προς πλεονέκτημα της Ουκρανίας και ήταν μειονέκτημα για τον Κρεμλίνο λόγω κυρώσεων. Και δεν μπορώ να πω ότι όσο παραμένουν κυρώσεις ότι είναι αρνητικά τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Και κάτι που θα πω το οποίο ενδεχομένως ε, να προκαλέσει αντιδράσεις. Ναι, η επίσημη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι υποχρεώσεις της ΜΕΝΣ και είναι να ε, εφαρμοστούν και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία. Αλλά νομίζω ότι τις συζητήσεις που έκανα αναγνωρίζουν οι ηγέτες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης πως επειδή είναι οθήτης η Ρωσία θα πρέπει πρώτα η Ρωσία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της. Και για το λόγο αυτό παρόλο που έχουμε αρκετά κακούς όρους συμφωνία αυτή. Η εφαρμογή που έγινε και η διαδικασία της Μίσκ, του Μίνσκ δεν ήταν τελικά αρνητική. Δεν έχει ε, οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, γιατί έχουμε κάθε μέρα παραβιάσεις. Οι περισσότερες γίνονται από τη ρωσική πλευρά του μετόπου. Πιστεύω όμως πως η συμφωνία αυτή είναι ικανοποιητική για όλους, ε, τους βολεύει όλους, οπότε το επόμενο εξάμεινο δεν θα καταληθεί για την τάξη, τη μεταψυχροπολεμική τάξη. Ναι, ήταν οι ηγέτες της ε, Σοβιετικής Ένωσης που αποφάσισαν να την καταλήξουν. Γιατί, γιατί πια είχε εξαντληθεί. Και ήταν σημαντικό να καταληθεί με ειρηνικό τρόπο, αλλά επειδή έγινε πραγματικότητα αυτές οι παγωμένες σειράξεις από τη στιγμή που εξαφανίστηκε η Σοβιετική Ένωση, ε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να πείτε ότι ήταν η βία, η πλευρά της κατάλυσης και επειδή είναι ανοιχτά ρεβιζιονιστής ο κύριος Πούτιν, αυτό γίνεται όλο και οξύτερο. Και βέβαια είναι και πιο δυνηρή η κατάσταση στη Γεωργία, εκτός από τα όσα συνέβησαν με την Ουκρανία. Η θέση μου είναι πως θα πρέπει να ενισχύσουμε τις κυρώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι το επιθυμεί η Ευρώπη. Και για την περίπτωση και την ανάλυση που έκανε ο κύριος Χοντορκόφσκι, έχει δίκιο. Στη Ρωσία θεωρούν πως οι κυρώσεις δεν είναι κατά του Κρεμλίνου αλλά κατά των Ρώσων. Και θα ήταν πολύ δύσκολο για μας, δεδομένων ε, των φημωμένων ε, ΜΜΕ στη Ρωσία, ε, να αλλάξουμε αυτή την ε, άποψη. Αλλά μπορούμε να προωθήσουμε τη συζήτηση προς σωστή κατεύθυνση ενδεχομένως. Σίγουρα οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών γνωρίζουν πού βρίσκονται τα δισεκατομμύρια του κυρίου Πούτιν μένα στη Δύση. Και αυτό νομίζω πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε. Sure that the... Our... Και όχι μόνο να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά να εξασφαλίσουμε πως οι πληροφορίες αυτές το εκπέμπουν ε, και στη Ρωσία έτσι ώστε να ξέρουν οι Ρώσοι που έχει στείλει τα λεφτά του ο κύριος Πούτιν και η συμβολή του βέβαια, όχι μόνο ο ίδιος. κύριο Ρογκοζίν, για παράδειγμα, έχει δισεκατομμύρια στη Δύση, δεν το ξέρω. Αλλά έχουμε τον κύριο Σέτσιν που έχει χρήματα στη Δύση και όλα αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια έτσι ώστε να το γνωρίσουν και οι Ρώσοι. Και να ξέρουμε και ποια είναι τα μέλη οικογενειών των αξιωματούχων του Κρεμλίνου που ζουν στη Δύση. Δεν χρειάζεται να δώσουμε διευθύνσει, να του πούμε πού ζουν, σε ποιε χώρες. Οπότε, όταν οι υπερπατριώτες στη Μόσχα μιλάνε για την παρεκμασμένη Δύση, να γνωρίζουν πως οι ηγέτες αυτές στην πραγματικότητα περνάνε καλά στη Δύση. Ναι, είμαι σκεπτικιστής για το πόσο καταλαβαίνει την Ρωσία ο κύριο Τραμπ. Δεν γνωρίζω όμως αν τα όσα είπε στην εκστρατεία θα αποτελέσουν κομμάτι ιστορικό της εκστρατείας ή αν θα γίνουν κομμάτι της ε, αμερικανικής πολιτικής. Δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα, γιατί οι σύμβουλοι τους δεν μοιάζουν να έχουν τις ίδιες απόψεις, παρόλο που ε, στην αίθουσα ε, επιγόντων περιστατικών θα έχουμε και άλλες απόψεις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλές πολιτικές τέτοιες που να προχωρούν σε ενθάρρυνση του κυρίου Πούτιν. Θα ήταν κακή πολιτική του κύριου Τραμπ να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί καμία από αυτές τις πολιτικές δεν θα τον κάνει πιο δημοφιλή οι πιο πετυχημένους στον Αμερικανικό λαό και χρειάζεται να τον στηρίξει και το Κογκρέσο για να συνεχίσει με πολιτικές που θα τον κάνουν πετυχημένο και δημοφιλή. Και τέλος, αν παρόλα αυτά ακολουθήσει τη λάθος κατεύθυνση, νομίζω ότι οι ψηλά ιστάμενοι, ή μάλλον οι μεγάλες ε, πολιτικές φυσιογνωμίες από το Κογκρέσο θα του ε, αντιταχθούν τώρα. Άκουσα τι είπε ο κ. Σακιασβίλη και εγώ. Η κλεπτοκρατία αυτή ήταν πρόβλημα όχι μόνο για την Ουκρανία και για τη Μόσχα και για τα υπόλοιπα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και θεωρώ πως έχει γίνει σοβαρή μεταρρύθμιση στην Ουκρανία, όχι πάντα υπό την ηγεσία της κυβέρνησης και κάποιες φορές ενδεχομένως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και ε, το Διεθνές και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν επιβάλει μεταρρυθμίσεις για να προσφέρουν ε, βοήθεια. Ακούσαμε για την αιρεσιμότητα. Οπότε σύσταση δική μου είναι μια σκληρή αγάπη με προϋποθέσεις τη μεταρρύθμιση, με περισσότερα κονδύλια και μαζί με αυτή τη σκληρή αγάπη και τη μεταρρυθμίση που είδαμε στην Ουκρανία και αυτές τις φοβερές ηλεκτρονικές δηλώσεις που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες ε, να καταφέρουμε τη διαφθορά αυτή να την περιορίσουμε. Δεν μπορούμε να την πατάξουμε πλήρως, αλλά να την περιορίσουμε. Και να αυξήσουμε τα κονδύλια που στέλνουμε στον Ουκρανικό λαό. Αυτό ήθελα να σας συστήσω. Και τέλος, τι έγινε την τελευταία δεκαετία. Ήταν δυνατή η Δύση. Ήταν αρκετά γρήγορη αντιδράσεις Όχι καθυστερήσαμε, ήμασταν αδύναμοι. Αν είχαμε ε, αντιδράσει σωστά στη Γεωργία θα είχαμε αποφύγει την Κρυμαία και αν είχαμε αντιδράσει για την Κρυμαία θα είχαμε αποφύγει τον Τον Μπάς. Οπότε νομίζω ότι δεν δείξαμε πυγμή τα τελευταία δέκα χρόνια. Είμαστε σε άσχημη θέση σήμερα. Ήμουν πολύ επικριτικός ε, στη σύνοδο του, της Ουαλίας όταν μας είπαν ότι το ISIS είναι υπαρξιακό πρόβλημα για το ίδιο το ΝΑΤΟ. Όχι, αυτό είναι αστείο, όχι για τη συμμαχία, για κάποια κράτη. Αλλά μία ανεξέλεγκτη πυρηνική δύναμη που έχει την ισχύ της ε, Ρωσίας, ναι, είναι απειλή για τη συμμαχία και το ότι δεν το αναγνωρίσαμε αυτό στην Ουαλία ήταν αποτυχία. Το αναγνωρίσαμε στη Βαρσοβία και πιστεύω πως αν δεν είχαμε τις πρόσφατες εκλογές στη ΣΥΠΑ, κάποια φαινόμενα τα οποία διαπιστώσαμε πρόσφατα να λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία, θα μας ανησυχούσαν περισσότερο. Πάντως, εγώ για την Αμερικανική πολιτική σκηνή είμαι τελικά αισιόδοξο και πιστεύω πως θα καταφέρουμε να δούμε και στη Γαλλία τα πράγματα να πάνε να ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Θα το πω αυτό αργότερα. Εξοχότατε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνεδρίαση. Αρχικά ε, θα ήθελα εγκάρδια να ευχαριστήσω όλους τους διερμηνείς ε, για την ε, δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 8 Δεκεμβρίου πρωί στις 9 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.